Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε, η ιδέα που είχαμε στην αρχή να αναβάλουμε για λίγο την έναρξη της συνεδρίασής μας από τις 3 στις 3 και 10 ήταν μια εξαιρετική ιδέα. Διότι όπως βλέπετε έχουμε εδώ πέρα πολύ περισσότερους συναδέλφους και μπορώ να σας πω ότι στις 3 μόνο 5 ήμασταν εδώ. Μόνο πέντε ευρωβουλευτέ. ήταν εδώ παρόντες στην αίθουσα. Οπότε, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Είναι η πρώτη μέρα εργασιών μετά τις θερινές διακοπές εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Έχουμε τις ακροάσεις που έρχονται όπου να είναι με τους υποψηφίους επιτρόπους για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε να ετοιμάσουμε και, την, και συναντήσεις με τους επιτρόπους, την Ελικρού, τον Έτιγκερ, την κυρία Κουίν, που είναι τώρα επίτροποι, γιατί θέλουμε να μας ενημερώσουν για τις τρέχουσες δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε και τις ακράσεις, όπως σας είπα. Θα αρχίσουν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ήδη την επόμενη εβδομάδα εμείς ως Επιτροπή Ήτρε πρέπει να ετοιμάσουμε τρεις ερωτήσεις προς κάθε υποψήφιο επίτροπο ο οποίος θα έρθει στην Επιτροπή μας. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα πότε θα τους δώσουμε τις ερωτήσεις κτλ. Πάντως θα αποφασιστεί ο πλήρης ε, κατάλογος των υποψηφίων επιτρόπων τώρα στα μέσα αυτής της εβδομάδας Μέχρι τη Δευτέρα το πολύ την επόμενη θα έχουμε όλο τον κατάλογο. Λοιπόν, όπως σας είπα έχουμε πολλή δουλειά που μας περιμένει. Ας μην μακρηγορούμε λοιπόν. Για τις καλοκαιρινές διακοπές θα τα πούμε ιδιαίτερος μετά τη συνεδρίαση. Ας έρθουμε λοιπόν στην ημερήσια διάταξη, την έχετε στους φακέλους σας όλοι. Αν δεν υπάρχουν σχόλια, παρατηρήσεις, συμφωνούμε ότι εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Θέλω επίσης να λάβετε υπόψη σας ότι το σημείο 16 είναι τα διάφορα. Οπότε στα διάφορα μπορείτε να θέσετε ό,τι νομίζετε. Σημείο δεύτερον, έγκριση των πρακτικών. Πρόκειται βέβαια για την ε, τη συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής μας που είχαμε στις 7 Ιουλίου. Έχετε και τα πρακτικά αυτά στους φακέλους σας. Τα πρακτικά θεωρούνται εγκεκριμένα εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Ωραία, περνάμε λοιπόν στο τρίτο σημείο στην ημερήσια διάταξη, ανακοινώσει του Πρόεδρου. Δεν θα λάβει χώρα συνεδρίαση των συντονιστών σήμερα. Συνεπώς, στο σημείο 15 που αφορά την διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές που προβλέπεται να λάβει χώρα στη Λίμα στο Περού, 1 με 12 Δεκεμβρίου του 2014, θα λάβει χώρα σήμερα. Η συζήτηση για το θέμα αυτό δηλαδή σήμερα, μετά το σημείο 6 θα περάσουμε στο σημείο 15, αφού δεν θα συνεδριάσουν οι συντονιστές σήμερα. Θα συζητήσουμε λοιπόν για τη διάσκεψη αυτή όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές και θα ανταλλάξουμε απόψεις. Βέβαια η ένβη τελικά θα αποφασίσει. Εμείς πρέπει να ετοιμάσουμε τη γνωμοδότησή μας για την ένβη. Αυτά όσον αφορά αλλαγέ στην ημερήσια διάταξη. Περνάμε τώρα στο σημείο 4. Γενικό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το Οικονομικό του 2015, όλα τα τμήματα. Εδώ επιτρέψτε μου να σας πω δύο λόγια για αυτό το θέμα εγώ. Πρώτα απ' όλα επί της διαδικασίας. Όπως γνωρίζετε η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών όσον αφορά τις γραμμές του προπολογισμού ήταν 19 Αυγούστου 2014. Υποβλήθηκαν 161 τροπολογίες. Βέβαια πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι ήταν μεγάλη τιμή για μένα που με ορίσατε εισηγητή για αυτό το θέμα. Για τον προπολογισμό του 2015. Μεγάλη τιμή για μένα να αναλάβω την ευθύνη αυτή από πλευράς της Επιτροπής και των Συντονιστών. Ευχαριστώ επίσης και τους σκιώδεις εισηγητές και όλους τους ευρωβουλευτές που επέβαλαν τροπολογίες. Ε, κυρίως επειδή χρειάστηκε να δουλέψουν κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών. Τα καταφέραμε όμως νομίζω. Μπορώ λοιπόν να υποστηρίξω τις περισσότερες από τις τροπολογίες σας. Μάλιστα έχω ετοιμάσει και 94 τροπολογίες εγώ ίδιος, που μοιάζουν πάρα πολύ με αντίστοιχες δικές σας. Άρα συμφωνούμε μεταξύ μας. Έρχομαι τώρα στο περιεχόμενο του σχεδίου γνωμοδότησης που ετοίμασα. Όπως είπα, ε, τον, και τον Ιούλιο, πιστεύω ότι οι περικοπές που έκανε το Συμβούλιο στο σχέδιο προπολογισμού που πέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2015 είναι δικαιολόγητες. Είναι το πιο βασικό και βαρισίμαντο που περιλαμβάνει η γνωμοδότησή μου. Πραγματικά ανησυχώ ιδιαίτερα για τις περικοπές αυτές που έχει επιφέρει το Συμβούλιο, ιδιαίτερα σε τομείς όπως είναι η καινοτομία, η έρευνα, οι υποδομές, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η ενέργεια. Ήδη τώρα δεν έχουμε αρκετά χρήματα στον ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό τώρα που μιλάμε για να γίνουν οι πληρωμές που πρέπει να γίνουν. Άρα οι περικοπές που προτείνονται θα επιδεινώσουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση πολιτή προγράμματα όπως είναι ορίζοντας 2020, το Κόσμε, η διευκόλυνση για τη σύνδεση στην Ευρώπη. Είναι όλα αυτά επιτεύγματα και στόχοι που έχουμε για την Ευρώπη το 2020. Πράγματα πολύ σημαντικά για μας και που αποφασίστηκαν πριν από δύο χρόνια ήδη. Ο προπολογισμό λοιπόν του 2015, μια που όλα αυτά τα θέματα μόλις ξεκινάνε, ο προπολογισμό του 2015 πρέπει να φροντίσει να υπάρξει η αναγκαία πρικοδότηση για να μπορέσουν και να συνεχιστούν οι πρωτοβουλίες αυτές. Χρειάζεται ε, πολύ στενό συντονισμό μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρών μελών και περιφερειών. Είναι κάτι αναγκαίο. Και θα σας δώσω και ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Καινοτομία και την Τεχνολογία. Εμείς έχουμε την ευθύνη για το Ινστιτούτο αυτό. Έτσι αποφασίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αποφασίστηκε δηλαδή να δημιουργηθεί το Ινστιτούτο αυτό, όπως επίσης και διάφοροι εκτελεστικοί φορείς. Πρέπει να έχουν τα χρήματα που χρειάζονται για να φέρουν σε πέρα τις αρμοδιότητες που έχουν αναλάβει. Αυτό όμως δεν είναι δυνατόν με τον προπολογισμό αυτόν. Συνεπώς, έτσι με αυτή τη σύντομη εισαγωγή, τις σύντομες αυτές παρατηρήσεις, θα ήθελα να ζητήσω από τους κοιόδης εισηγητές να πάρουν το λόγο και τους συντονιστές. Αν θέλετε, παρακαλώ. Αλλά να είσαστε Σύντομη, δύο λεπτά ο καθένας θα έλεγα. Γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και μετά και οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές, αν θέλουν, μπορούν ένα λεπτό ο καθένας να μας μεταφέρουν τις παρατηρήσεις τους. Αρχίζει η συζήτηση από το ΕΛΚ. Ποιος θα ήθελε να πει κάτι. Κανείς από το ΕΛΚ. Α, παρακαλώ. Κύριε Δεν έχω τίποτα να προσθέσω σε όλα αυτά τα πολύ σωστά που είπε ο Πρόεδρος. Θέλω απλά να πω ότι όσον αφορά τα πολυετή προγράμματα στο γεγονός ότι υπάρχει ελλειπής ε, χρηματοδότηση, το θέμα δεν είναι μόνο ότι πράγματι υπάρχει η ελλειπής αυτή χρηματοδότηση, αλλά και το εξής πρόβλημα, ότι τα αναβάλουμε συνεχώς τα προγράμματα και έτσι γίνονται και τα δαπανηρότερα. Αυτό αποδείχθηκε ας πούμε, στο πρόγραμμα COSME ή αν θέλετε στην πυρηνική σύνδεξη ε, Λόγω ακριβώς αυτής της ε, οικονομικής διαχείρισης που κάναμε που οδήγησε συνεχώς σε υποχρηματοδότηση τελικά καταλήξαμε, που σας είπα, σε υψηλότερο κόστος και θα ήταν πολύ καλύτερα από την αρχή να είχαμε επιλέξει διαφορετική λύση. Άρα δηλαδή η δική μου παράκληση είναι όχι μόνο να εξετάσουμε τον προπολογισμό του 2015, αλλά και να δούμε ποιο είναι αυτό το επιπρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της συνεχούς υποχρηματοδότησης στις γραμμές του προπολογισμού. Σας επαναλαμβάνω, ε, τα πολιτή προγράμματα κατέστησαν ιδιαίτερα δαπανηρά, οι ε, διαγωνισμοί, η προκήρυξη αγωνισμών επίσης. Άρα δηλαδή θα πρέπει να ζητήσουμε μια νέα βάση συνεργασίας ε, με την Επιτροπή Προεπολογισμών. Να μην περιοριζόμαστε μόνο στις αυστηρές μας αρμοδιότητες των ε, προϋπολογισμό, αλλά να συνεργαζόμαστε και σε άλλα θέματα με θέματα Επιτροπής Προϋπολογισμών. Γιατί στη δική μας την Επιτροπή μιλάμε για ένα κόστος της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ορισμένα προγράμματα θα υποστούν ζημιές, ε, πραγματικά είναι υποχρηματοδοτούμενα και εάν τελικά εκτελεστούν θα κοστίσουν πολύ περισσότερο και μόνο αυτό, αλλά ενδέχεται και να μην υλοποιηθούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιο ε, από κάποια άλλη πολιτική ομάδα να λάβει το λόγο. Ο κύριος Ρόιλ που είναι από την ίδια πολιτική ομάδα. Παρακαλώ πολύ, έχετε το λόγο. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να υποστηρίξω αυτά που ήδη είπε ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι είναι σημαντικό ως ε, Επιτροπή Βιομηχανίας και που ασχολείται με θέματα ε, προκαταβολών να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα ότι δεν συμφωνούμε, ότι αυτή είναι μια σαφής ε, λανθασμένη κατεύθυνση. Από το πρωί στο βράδυ ακούμε από όλες τις σημαντικές πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη ότι πρέπει να ασχοληθούμε με την ανάπτυξη, με την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τελικά Κανείς δεν σκέφτεται τίποτα άλλο από το να αναζητά τη λύση στην εκταμείευση περισσότερων κονδυλίων. Το θέμα όμως είναι τα κονδύλια να εκταμιεύονται για σωστό σκοπό και όχι όπως γίνεται τώρα. Οφείλουμε να στηρίξουμε την ε, βιομηχανική πολιτική, την πολιτική έρευνας. Ο κύριος ε, Νίλερ έχει δίκιο. Ε, πράγματι, αν δεν δει κανείς αυτή τη μακριά λυσίδα και τις ε, συνέπειες μιας λανθασμένης απόφασης, ε, τότε προκύπτουν πάρα πολλά προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Πρόεδρε, εμείς στηρίζουμε ανεπιθύλακτα αυτή την πρόταση και προτείνουμε επίσης ε, να ζητήσουμε την υποστήριξη συναντέλφων και να ζητήσουμε οπωσδήποτε και αλλαγές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Ταμποράνο. Πρόεδρε, εμείς ε, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά τα κονδύλια για την έρευνα και την ε, τεχνολογική ανανέωση, διότι τώρα πλέον είμαστε σε μία ήπειρο που θεωρείται ευημερούσα και δεν πρέπει να θυσιάσουμε τίποτα απολύτως. Υπάρχουν πάρα πολλά παράδοξα στοιχεία στην ε, λιτότητα. Πολλοί λένε ότι θέλουν να ανάπτυξη και θέση απασχόληση, όμως είναι ακριβώς αυτές οι χώρες οι οποίες προκύπτουν δικαιολόγητες περικοπές. Γι' αυτό λοιπόν, λοιπόν εγώ στηρίζω αυτά που λέει ο συγητής και θέλουμε να στηρίξουμε όλες εκείνες τις τροπολογίες οι οποίες φαίνουν τον προϋπολογισμό στην αρχική του μορφή πριν από τις ε, περικοπές ε, του Συμβουλίου. Δεν πρέπει να γίνονται περικοπές για να χρηματοδοτούνται εξοπλισμοί και άλλα παρεμφερή προγράμματα. Ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος αλλά μιλήσατε πολύ περισσότερο από δύο λεπτά και έχουν ζητήσει το λόγο 11 συνάδελφοι. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Σωρίνο εκ μέρους των συντονιστών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους των ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα ήθελα να σας εκφράσω και τις δικές μας τις ανησυχίες όσον αφορά την ε, μη ε, επαρκή χρηματοδότηση, την πρόβλεψη επαρκών κονδυλίων για αυτό τον προπολογισμό. Διότι προβλέπετε περικοπή των κονδυλίων κατά περίπου 2%. Και αυτό αφορά στα κονδύλια τα οποία είναι απαραίτητα για να εφαρμοστούν προγράμματα. Προβλέπεται επίσης και περικοπή κατά 8,6% στις πληρωμές. Αυτό όμως είναι απαράδεκτο και κυρίως θέλω να πω ότι οι περικοπές βρίσκονται σε αντίφαση με αυτά τα οποία αναφέρθηκαν, ε, δηλώθηκαν αυτή την εβδομάδα. Ε, μάλιστα προχθές στη συνέντευξη κορυφής αποφασίστηκε ότι στις 7 Οκτωβρίου θα εξεταστούν εντελεχώς όλα αυτά τα θέματα. Αυτό είναι η μία αντίφαση και η δεύτερη αντίφαση είναι σε αυτά που πρότεινε ο πρόεδρος Κομισιόν, ο κύριος Γιούγκερ, ο οποίος μίλησε για ευρωπαϊκό ε, πρόγραμμα απασχόλησης και τεχνολογίας που θα ασχοληθεί με θέματα ενέργειας, με νέους βιομηχανικούς κλάδους και με την εφαρμοσμένη έρευνα. Αυτό από μόνο του είναι οξύμορο. Υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις και αυτό κοστίζει πάρα πολύ τόσο σε θεσμικό όσο και σε δημοκρατικό επίπεδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενος ε, συντονιστής, ο κύριος Σιλικιώτης παρακαλώ. Ε, θα μιλήσει ο συνάδελφος από την ΚΟΕ, εκ μέρους της ΚΟΕ, Ζωάο Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μην ε, υπολογίσετε αυτά τα 20 δευτερόλεπτα του αδελφέ, ήθελα στη διάθεση, στο, ε, στο χρόνο που έχω να αναφερθώ σε τρία στοιχεία. Κάντε ένα απολογισμό. Πρώτα απ' όλα, συμφωνούμε με την κριτική που ασκείται στο Συμβούλιο. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση, πράγματι. Οι χώρε αυτέ ακριβώ οι οποίε ήθελαν να επιβάλλουν αυτόν τον προπολογισμό σε άλλες χώρες, τώρα θέτουν υπό την εφαρμογή του, την υλοποίηση αυτή, αυτού του έκτακτου προπολογισμού. Γι' αυτό εμείς είμαστε κατά αυτών των εγκάρσιων περικοπών που προτείνει το Συμβούλιο. Δεύτερον, πολύ γρήγορα, θα ήθελα να πω ότι δύο είναι οι σημαντικές ανησυχίες που εκφράζονται και με τις τροπολογίες της ομάδας μας. Πρώτα απ' όλα ό,τι αφορά το πρόγραμμα Horizon 2020. Παρά την ενίσχυσή του, το πρόγραμμα αυτό δεν ε, την χάνει δίκες μεταχείρισης, διότι λίγες είναι οι χώρες οι οποίες απορροφούν το μεγαλύτερο τμήμα των κονδυλίων. Έπρεπε λοιπόν και εν μέρει επιτεύχθη αυτό να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα αυτό και η συνοχή με την εισαγωγή μιας κατηγορίας για την αριστεία και την αύξηση της συμμετοχής. Πιστεύουμε ότι τα κονδύλια είναι ανεπαρκή στο κομμάτι αυτό και δεν μπορούν ε, να προωθήσουν ούτε να έχουμε καλύτερη διαχείριση, ούτε να έχουμε μεγαλύτερη συνοχή στο πρόγραμμα πλαίσιο. Θέλουμε λοιπόν αυτή η κατηγορία να ενισχυθεί σημαντικά. Ταυτόχρονα είπαμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά και το έργο των ΜΜΕ. Στην πράξη βλέπουμε ότι πολύ λίγη είναι η πρόσβαση που έχουν στα κοινοτικά κονδύλια ΜΜΕ και έχουμε καταθέσει διάφορες προτάσεις τροπολογίας, τροπολογιών ώστε να ενισχυθούν ε, τα κονδύλια που προορίζονται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για να είναι καλύτερη η πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, σε δάνεια, σε ενισχύσεις. Επίσης βλέπουμε με λύπη μας ε, ότι εσείς απορρίπτετε όλες τις προτάσεις τροπλής της ομάδας μας. Για τους πρασίνους παρακαλώ τώρα. Πρώτα απ' όλα, λέει ο κύριος Τούρμες, ε, ελπίζω να περάσατε όλοι πολύ καλές διακοπές. Εκπροσωπώ τον κύριο Μπουτικόφερ, που ήταν ο σκιώδης για την ομάδα μας. Εκπράσουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας και πρέπει να καταπολεμήσουμε το Συμβούλιο όλοι μαζί από κοινού είναι απαράδεκτη στάση του και ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Κατά δεύτερον, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει όλοι να στηρίξουμε τις προτάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε χάρη στον Αντώνιο Ταγιάννη το πρόγραμμα COSME, η Κομισιόν πρότεινε, υποσχέθηκε θα 3 δις για τις ΜΜΕ Φτάνω μέχρι το 2020 και αυτό που προτείνει για το 2014-2015 η Κομισιόν ε, δεν εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο της ε, σταδιακής αύξησης. Είναι υπολοιπό, υπολείπονται τα ποσά αυτών που είχαν ε, προταθεί αρχικά. Τώρα τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε τι γίνεται με τα παιχνίδια στην ενέργεια με τον κύριο Πούτιν, ενεργειακή απόδοση και τα σχετικά με την ενέργεια γενικά είναι ίσως πιο σημαντικά από ποτέ θέματα για μας. Θα θέλαμε λοιπόν ιδίω για τα προγράμματα ενεργειακής απόδοσης ε, να δοθεί μεγαλύτερη ενίσχυση ε, οικονομική. Έχουμε επίσης το ΙΤΕΡ ε, ή το Γκαλιλαίο για προγράμματα για τα οποία εμείς εκφράζουμε έντονες επιφυλάξεις, διότι δεν νομίζουμε ότι αποδίδουν αυτά τα προγράμματα Το Γαλιλαίο έχει ε, και το εξή μειονέκτημα για τους νέους συνάδελφους το λέω πριν από 10 χρόνια μας το πλάσαραν τον Γαλιλαίο ως ένα πρόγραμμα το οποίο θα χρειαστεί μηδέν δημόσια χρηματοδότηση τώρα που βρισκόμαστε πόσα δις απαιτούνται και βλέπουμε ότι δεν μπαίνει και σε τροχιά το όλο πρόγραμμα τελικά και για το ίτερ σε 50 χρόνια. Από το 1950 που είχε δοθεί υπόσχεση μέχρι το 2000 ότι θα έχουμε δωρεάν ενέργεια, τώρα που θα φτάσουμε το 2080. Κατά λοιπόν είμαστε ως ομάδα αυτών των δύο προγραμμάτων. Για φανταστείτε ότι οι μεγαλύτεροι εγκέφαλοι, τα μεγαλύτερα μυαλά λένε ότι πρέπει να αυξηθεί η ενεργική απόδοση και όχι να δαπανούμε χρήματα και χρόνο με αυτά τα προγράμματα, τα άχρηστα. Πρόεδρος, κύριος Πέντερσεν τώρα και επειδή έχω δέκα ε, συναδέλφου στον κατάλογο θα μειώσω το χρόνο στο ένα λεπτό. Κύριος Πέτρισεν, είναι άδικο κύριε Πρόεδρε αυτό, γιατί οι ε, μίλησαν πολύ περισσότερο διορθώνω, ήταν είτε συντονιστές είτε σκιώδεις οι προηγούμενοι. Και αυτοί είχαν δύο λεπτά στη διάθεσή τους, τώρα οι υπόλοιποι ένα λεπτό. Για να το πω πιο ξεκάθαρα. Κύριος Πέτρισεν, θα είμαι πολύ σύντομος. Η Άλντε συμμερίζεται μεγάλο μέρος των απόψεων που διατυπώθηκαν μέχρι τώρα συμφωνούμε και με ένα μεγάλο μέρος της ανάλυσης και των δυσκολίων που αντιμετωπίζουμε. Εκ μέρους λοιπόν της ομάδας ALDE, θέλω να πω ότι εμείς θα ψηφίσουμε υπέρ της ε, ε αποκατάστασης του προϋποσμού στα αρχικά του επίπεδα, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και προσβλέπω στις μελλοντικέ συζητήσεις. Πρώτα, σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκροστέτ έχει τώρα το λόγο. Ε, κύριε Πρόεδρε, τι μπορούμε να, να πούμε. Λέμε ότι πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη στην Ευρώπη. Πώς το λέμε αυτό και από την άλλη μειώνουμε τον προπολογισμό που στόχο έχει ακριβώς να ε, οδηγήσει σε ανάπτυξη. Και αποθαρρύνουμε και πιθανούς επενδυτές. Θα πρέπει η δημοσιονομική στήριξη προς τις ΜΜΕ να συνεχιστεί, αυτή η χρωματοδοτική στήριξη προς τις ΜΜΕ και προς όλους τους στρατηγικούς τομείς, όπως ε, της ενέργειας θα πρέπει ο προϋπολογισμός να παραμείνει στα ευκταία επίπεδα. Αυτό είναι σημαντικό γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχει καμία συνέπεια στην πολιτική μας και πόσο μάλλον θα χάσουμε, θα απολέσουμε εντελώ την αξιοπιστία μας. Ευχαριστώ. Από ό,τι ξέρω, το 3% του ΑΕΠ δεσμεύτηκαν όλοι οι κρατών και κυβερνήσεων να δαπανούν για την ενέργεια και για την έρευνα και ανάπτυξη μας συγκεκριμένα. Δεν το κάνουν όμως. Μιλάμε ε, για αυτό τον προπολογισμό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ε, υπάρχουν επαρκείς δαπάνες για τις κατηγορίες αυτές. Ζητούμε λοιπόν από τι εθνικέ κυβερνήσει ε, να τηρήσουν τι δεσμεύσει του. Děkuji, pane předsedo. Já το Συμφωνώ με τα όσα μόλις είπε ο καθηγητής Σέγκελ. Γνωρίζουμε τη δημοσιονομική κατάσταση που είναι αρκετά ζωφερή, δεν υπάρχουν κονδύλια. Στην προκειμένη περίπτωση όμως θα πρέπει να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητές μας. Κατά το παρελθόν πολύ λόγος έγινε για αυτές τις προτεραιότητες και νομίζω ότι συμφωνήσαμε οι περισσότεροι στην έρευνα και ανάπτυξη ως προτεραιότητα. Όπως είπατε, δεν πρέπει να επιτρέψουμε αυτές τις περικοπές, ιδίως ε, για προγράμματα τα οποία έχουν ήδη εκκινήσει. Με τον Κλό όμως πρέπει να διαφωνήσω. Νομίζω ότι το πρόγραμμα Γκαλιλαίο πρέπει να περατωθεί και είναι μία από τις προτεραιότητες δεν μπορεί αυτό το πρόγραμμα να εφαρμοστεί μεμονωμένα από καμία ευρωπαϊκή χώρα. Πρέπει να γίνει κοινή προσπάθεια. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε την επαρκή χρηματοδότηση στην έρευνα και την ανάπτυξη. Αντιπρόεδρος. Όσοι ήταν εδώ στην προηγούμενη θητεία, σε αυτούς θέλω να πω, αλλά και στους καινούριου κυρίως, το πόσο δύσκολο ήταν να φτάσουμε σε αυτό το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δύσκολο για μας, ε, προφανώς και ο προϋπολογισμός δεν μας ε, ικανοποιούσε και προσπαθήσαμε να βρούμε ένα συμβασμό. Ο κύριος ε, Λαμασούρ είχε ασκήσει ιδιαίτερη κριτική και εμείς θέλαμε πολλά περισσότερα κονδύλια για το πρόγραμμα Ορίζοντας που ήταν αυξημένο ο προπολογισμό του από τον προηγούμενο αλλά θέλαμε ακόμα περισσότερα. Και τελικά δεχθήκαμε ένα συγκεκριμένο ποσό διότι υπήρχε αυτό το περίφημο front loading ή εμπροστοβαρής χρηματοδότηση και ε, σε αυτό το πλαίσιο της εμπροστοβαρής χρηματοδότησης ε, είχαμε στην αρχή περισσότερα κονδύλια και αργότερα ε, θα υπήρχε μείωση. Αν όμως τα ακυρώσουμε όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι ο δρόμος θα είναι πάρα πολύ δύσκολος και Θέλω επίσης να προσθέσω και δύο άλλα πράγματα. Πρώτον, όσον αφορά το πρόγραμμα COSME, αυτό θα αυξηθεί γιατί είναι πολύ σημαντικό και το ΕΑΖΙ που αφορά τις ε, κοινωνικές πολιτικές ε, και αυτό έχει κυρίως σχέση και την πρόοδο της κοινωνίας σε σχέση με την τεχνολογία. Ευχαριστώ πολύ. αυτόν τον προπολογισμό μας ε, λείπουν ε, τα κονδύλια και έτσι λοιπόν ε, αν δεν υπάρξει αύξηση θα έχουμε διαρθρωτικά ελλείμματα. Κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα το πώς ακριβώς θα πείσουμε το Συμβουλίο να τηρήσει τις υποσχέσεις του. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό επιτέλους να τελειώσει αυτό το σύστημα των ιδίων πόρων για να αλλάξει και η κατάσταση και αυτό θεωρώ ότι είναι το βασικότερο καθήκον μας επόμενος η Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ρούτε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τέσσερα σημεία θέλω να αναφέρω και σας ευχαριστώ πολύ για την μέχρι τώρα συζήτηση που πηγαίνει προς την κατεύθυνση που σκεφτόμαστε κι εμείς. Το πρώτο μου σημείο έχει να κάνει με το Horizon 2020 για να σας πω ότι πράγματι όταν τώρα μάλλον που η Ευρώπη χρειάζεται τόσο πολύ επενδύσεις που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη, προγράμματα όπως είναι το Προγραμμά πλαίσιο, το Horizon, είναι αυτά που περισσότερο χρειάζονται για την έρευνα και την καινοτομία στην Ευρώπη. Αυτό είναι το πρώτο μου λοιπόν σημείο και να υπογραμμίσω επίσης ότι πάντα εμείς 100% τηρήσαμε τις υποχρώσεις μας. Δεύτερον, Όσον αφορά τις περικοπές από πλευράς του Συμβουλίου, θα έχετε διαπιστώσει ότι τα ποσοστά διαφέρουν. Αν μιλάμε για τον προπολογισμό της έρευνας, έχουμε περικοπές πάνω από 10%, ενώ σε άλλες γραμμές του προπολογισμού υπάρχει μείωση 0,1%. Οπότε διαπιστώνουμε ότι οι περικοπές που γίνονται στην έρευνα είναι πολύ πιο σημαντικές από ό,τι οι περικοπές που γίνονται αλλού. Τι σημαίνει αυτό για την εφαρμογή των δικών μας προγραμμάτων και για τη χρήση του προπολογισμού. Αυτό σημαίνει ότι φέτος εμείς στην έρευνα, στην Επιτροπή δεν θα μπορέσουμε να τηρήσουμε τις ευατικές μας υποχρεώσεις και να πληρώσουμε τους δικαιούχους όπως τους έχουμε υποσχεθεί. Το 2015 δεν θα έχουμε ακόμα περισσότερες δυσκολίες να τηρήσουμε τις βατικές μας υποχρεώσεις. Επιπλέον, αν δείτε τα τέλη των προγραμμάτων. Κάθε φορά μειώνεται ο προϋπολογισμός, που σημαίνει ότι μένουν ε, απλήρωτες υποχρεώσεις από το παρελθόν. Και στα τέλη του 2020 θα έχουμε κάπου 20% του ορίζον 2020 χωρίς να έχουν γίνει κανονικά οι Δηλαδή θα κουβαλάμε ένα χρέος επειδή κάθε χρόνο δεν θα πληρώνουμε και δεν θα τηρούμε τις υποχρεώσεις μας πλήρως. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, <clears throat> ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξή σας. Ειλικρινά δεν ε, βρήκα καμία διαφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων πρώτα απ' όλα για τα θέματα αυτά. Ίσως κάποιες μικρές αποχρώσεις, ναι εντάξει, μικρές. Αλλά όλοι μας θα θέλαμε... Καλά Κλόντ, έχεις δίκιο. Έλεγα λοιπόν ότι όλοι μας θέλουμε να επιστρέψουμε σε έναν μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Περισσότερα κονδύλια, κυρίως για την έρευνα και την καινοτομία, προκειμένου να έχουμε ανάπτυξη στην Ευρώπη. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με τα περισσότερα σημεία. Τώρα, δύο λόγια για το χρονοδιάγραμμα. Όπως γνωρίζετε, η διαδικασία όσον αφορά τον προπολογισμό 2015 χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι η γνωμοδότηση όσον αφορά τις τροπολογίες επί του προπολογισμού συζητάμε τις τροπολογίες και η γνωμοδότηση όσον αφορά το ψήφισμα για τον ε, προπολογισμό, την έκθεση μάλλον για τον προπολογισμό. Αύριο θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες, το πρώτο σκέλος δηλαδή. Αύριο, 2 Σεπτεμβρίου 2014. Προθεσμία τώρα για τις τροπολογίες όσον αφορά το σχέδιο προπολογισμού είναι 3η Σεπτεμβρίου 2014 στις 12 το μεσημέρι. θα ψηφίσουμε στην Ήτρε τη γνωμοδότηση στον προπολογισμό στις 25 Σεπτεμβρίου 2014. Σε τρεις εβδομάδες λίγο πολύ. Και θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια, στη δεύτερη Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Στο Στρασβούργο. Γιατί έχουμε δύο τον Οκτώβριο Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Οκτώβριος 2014 εννοείται. Αυτό είναι λοιπόν το χρονοδιάγραμμα και αύριο έτσι καλώς θα ψηφίσουμε ήδη τις τροπολογίες. Καλώς. Περνάμε στο επόμενο σημείο τώρα. Καλωσορίζω εδώ τον κύριο Γκόραν Μάρμπι, που είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σώματος Ρυθμιστών όσον αφορά τις επικοινωνίες. Πρόκειται για το BEREC έτσι ονομάζεται το σώμα αυτό. Πολύ σημαντικό όργανο όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες και την ψηφιακή ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι πολύ σημαντική η παρουσίαση αυτή. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που ήρθατε και θέλω να σας δώσω το λόγο για την παρουσίασή σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Προσπαθώ και εγώ να βρω την παρουσίασή μου, λέει ο μιλητής. Ηλεκτρονικά βέβαια την ψάχνω. Αρχίζω λέγοντά σα ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ και μεγάλη ικανοποίηση που μπορώ να σας παρουσιάσω την παρουσίαση αυτή. Πρέπει να σας πω ότι Θεωρούμε ότι εσείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είσαστε οι γονείς μας. Το Μπέρεκ βασίστηκε σε πρωτοβουλία της δικιάς σας Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν χρειάζεται εδώ να σας δώσω λεπτομέρειες για το τι έχω κάνει, να σας πω όμως ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ. Και αρχίζω την παρουσίασή μου τώρα. Υπάρχουν εδώ βέβαια και νέα μέλη που δεν ήταν στην προηγούμενη θητεία, γι' αυτό επιτρέψτε μου να κάνω μια σύντομη εισαγωγή για το ποιοι είμαστε και τι ακριβώς κάνουμε. Έχουμε 28 κρατη και είμαστε ρυθμιστές. Ίσως να μην είμαστε πιο δημοφιλείς. Πολύ συχνά λέμε ότι κανείς δεν είναι ευχαριστημένος με τη δικιά μας τη δουλειά. Γιατί, Γιατί εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βρούμε μια ισορροπία. Προσπαθούμε επίσης να λάβουμε υπόψη μας πάντα τις επιθυμίες των καταναλωτών και να κάνουμε τις σωστές επιλογές. Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές τα βάζουμε με τους φορείς των τηλεπικοινωνιών μέσα σε μια αγορά η οποία δημιουργεί μονοπόλια. Έχουμε και παρατηρητές, 8 κράτη-μέλη από υποψήφιες χώρες είναι και η Αλβανία μέσα σε αυτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης συμμετέχει. Ο ρόλος μας, και θα επανέλθω βέβαια σε αυτό πολλές φορές, είναι να είμαστε ε, ανεξάρτητοι ρυθμιστές των αγορών και να εξυπηρετούμε τους πολίτες. Εξαιτία όλων των χρηστών καταλαβαίνετε ότι η πρόκληση για μας είναι μεγάλη, γιατί όπως ήδη θα γνωρίζετε υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές στις τηλεπικοινωνίες, στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε ε, τις επικοινωνίες και έχουν αλλάξει πάρα πάρα πολλά πράγματα. Πριν από 10 χρόνια δεν υπήρχε το Skype, δεν υπήρχε το Facebook. Ο τρόπος επίσης που χρησιμοποιούμε τα πράγματα αυτά αλλάζουν και τη βιομηχανία Telecom αλλά και τις ρυθμίσεις. Τώρα, εσεί που ενδιαφέρεστε για το πώς δουλεύουμε, πρέπει να ξέρετε ότι δεν πρόκειται για ένα σώμα, πρόκειται για πολλά. Πρώτα απ' όλα έχουμε το Συμβούλιο Ρυθμιστών, 28 μέλη συν παρατηρητέ. Και επιπλέον έχουμε τη Διαχειριστική Επιτροπή, που ρόλος της είναι να ε, φροντίζει ότι φτάνει στα γραφεία στη Ρήγα, Μπέρεκ. Με 27 άτομα προσωπικό. Πώς δουλεύουμε λοιπόν. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους επικεφαλείς των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών. Μία από τις ιδιαιτερότητες που συζητούν πολύ είναι μα πώς δουλεύετε. Εσείς φτιάξατε ένα πολύ δημοκρατικό σύστημα βάσει του οποίου δουλεύει το ΠΕΡΚ. Εγώ λοιπόν έχω εκλεγεί για το 2014 και πριν από λίγους μήνες εκλέξαμε τον επόμενο πρόεδρο που θα είναι ο Φαντίμα Βαρός από την Πορτογαλία. Είναι εκ περιτροπής το σύστημα. Κάτι το οποίο δημιουργεί την ευκαιρία για πολλέ χώρε μέλη και η Σουηδία δεν είναι μια από τις πιο μεγάλες, αλλά παρόλα αυτά όλες οι χώρες, το διαπιστώνεται μέσα από μένα, όλες οι χώρες έχουν εξίσου τη δυνατότητα να βρεθούν επικεφαλής του διοικητικού αυτού συμβουλίου και να συζητούν επίσης ώρες με τους υπόλοιπους. Έχουμε ολομέλειες για να παίρνουμε αποφάσεις έχουμε και ένα δίκτυο επαφών με εμπειρογνώμονες που μας βοηθούν. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα που θα αρχίσει σύντομα είναι το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών μας. Και βασιζόμαστε και σε ομάδες εμπειρογνωμόνων. Τι μας ζητήσατε λοιπόν εσείς να κάνουμε. Πολύ απλά για να το πω, να αναρμονίσουμε κάπως τις ρυθμίσεις τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση, επειδή υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις χώρες μέλη. Έχουμε διαφορετικούς φορείς, έχουμε διαφορετικές, διαφορετική ζήτηση από τους καταναλωτές, διαφορετικές συνθήκες αγοράς, αλλά και διαφορετική νοοτροπία. Προσπαθούμε λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας το καλύτερο που υπάρχει σε κάθε χώρα και να το χρησιμοποιήσουμε. Στην τελευταία οικονομική κρίση είδαμε ότι πάρα πολλές επενδύσεις από τις χώρες μέλη, μάλλον πριν την κρίση, είδαμε πάρα πολλές επενδύσεις στον τομέα αυτό. Πολύ σημαντικό αυτό για τον οργανισμό μας. Κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι βοηθούμε τους εθνικούς ρυθμιστές. Σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Πάντως είμαι ευγνώμων για τη στήριξη που μας έχετε δώσει όλα αυτά τα χρόνια και για τις αποφάσεις που πήρατε εσείς στις αρχές της χρονιάς, εσείς εδώ στην Επιτροπή αυτή. Γίνονται πολλές συζητήσεις για την αναρμόνιση και για το πώς αυτή λειτουργεί στις χώρες μέλη. Είναι δύσκολο φυσικά να μετρήσει κανείς πόσο καλά κάνουμε τη δουλειά μας. Ένας τρόπος είναι η διαδικασία του άρθρου 7. Αυτό που συμβαίνει ότι με τις εθνικές αρχές και το έχω συζητήσει και με τους ευρωβουλευτές λέγοντας ότι είμαστε ανεξάρτητοι έτσι κι αλλιώς δεν ζητάμε από την κυβέρνησή μας κάθε φορά να, κάνουμε να πάρει κάποια απόφαση αλλά κάνουμε κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παίρνουμε λοιπόν πολλές αποφάσεις και η Μπέρεκ συμμετέχει στις ρυθμίσεις, παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν υπάρχουν σοβαρά διλήμματα, σοβαρές αμφιβολίες. Έτσι κι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την γνωμοδότηση της Μπέρεκ. Περισσότερες από τις κοινοποίησεις που πάνε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν να κάνουν με την εναρμόνιση. Λίγες φορές έχει σοβαρές αμφιβολίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάθε φορά που είχε τέτοιες αμφιβολίες αποσύρθηκαν οι εθνικοί ρυθμιστές. Τις περισσότερες φορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στηρίξει τη γνωμοδότηση της ΜΠΕΡΕΚ με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Μόνο σε πέντε περιπτώσεις από τις εκατοντάδες που έχουν φτάσει διαπιστώθηκε ότι η ΜΠΕΡΕΚ θεώρησε ότι ήταν αδικαιολόγητες οι σοβαρές αφιβολίες. Βέβαια εδώ μιλάω για στατιστικά δεδομένα, έτσι. Ποια είναι τα σημαντικά θέματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε το 2014. Η πρόταση για κανονισμό όσον αφορά τη συνδεδεμένη Ευρώπη και την ουδετερότητα των δικτύων αλλά και, και την περιαγωγή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από καιρό είχε ξεκινήσει με την πρότασή της, ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο τέλος. Όσον αφορά την ουδετερότητα δικτύων, υπάρχει κάτι σημαντικό. Κάθε φορά που εσείς μας ζητάτε να καταλήξουμε σε μία λύση, εμείς πιστεύουμε ότι το ανοιχτό δίκτυο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους Ευρωπαίους πολίτες. οι καταναλωτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν σωστά το διαδίκτυο με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Όσον αφορά την περιαγωγή, ξέρετε ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δικιά σας την πρόταση. Εμείς δουλεύουμε πάνω σε αυτό και προσπαθούμε να δούμε πώς θα εφαρμοστεί στο μέλλον. Παρακολουθούμε τη συζήτηση γιατί πιστεύουμε ότι η περιαγωγή είναι κάτι πολύ σημαντικό στην Ευρώπη. Κάτι άλλο που είναι όμως τεχνικό, αυτό είναι η σύσταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις σχετικές αγορές. Είναι όμως πολύ βασικό να δούμε πώς πιστεύουμε ότι θα εξελιχθεί η αγορά στο μέλλον. Αν δούμε τους διάφορους φορείς και αν δούμε ότι δεν χρησιμοποιείται πια τόσο πολύ φωνή, αλλά χρησιμοποιούνται τα ψηφιακά δεδομένα. Είναι μια σημαντική αλλαγή αυτή στην αγορά. Άρα και ο ορισμός για το πώς βλέπουμε τις αγορές στο μέλλον πρέπει να αλλάξει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν σε αρχές της χρονιάς έκανε μια σχετική πρόταση που εγκρίθηκε τον Ιούνιο από την Πέρεκ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως είναι εκείνη που την έκανε. Ε, πριν συζητούσατε για τον προπολογισμό, έτσι. Άρα έρχεται πολύ καλά αυτό που σας λέω τώρα. Λοιπόν, πώς θα πάει η Ευρώπη σε σχέση με άλλα σημεία του κόσμου. Πώς μπορούμε να μετρήσουμε την επιτυχία της Ευρώπης σε αυτό το τομέα. Κάποιες χώρες του κόσμου, πρέπει να σας πω, που είναι στην πρώτη γραμμή σε σχέση με τις λιπικοινωνίες είναι ευρωπαϊκές. Αλλά υπάρχει και το αντίθετο. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια πάντως. Στατιστικά μπορούμε να πούμε, και γι' αυτό σας δείχνω εδώ τη διαφάνεια, είναι γιατί η Μπέρεκ πιστεύει ότι έχουμε την επιλογή. Και εφόσον ο καταναλωτής έχει την επιλογή, υπάρχει ανταγωνισμός και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν σημαίνει ότι αν έχουμε το ευρωζωνικό, το σταθερό ή το κινητό, αυτή είναι όλη και όλη η επιλογή που έχουμε. Οι Ευρωπαίοι πολίτες πάντως έχουν πιο μεγάλη ταχύτητα για χαμηλότερο κόστος από ό,τι έχουν οι πολίτες της Ηνωμένες Πολιτείες δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν και άλλα τα οποία πρέπει να βελτιώσουμε. Συνεργαζόμαστε. Και είναι σημαντικό να συνεργαζόμαστε μαζί με εσά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να μπορέσουμε να επωφεληθούμε από την προηγμένη τεχνολογία που διαθέτουμε για να κάνουμε τα πράγματα ακόμα καλύτερα για τους Ευρωπαίου πολίτε. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μα είπατε και θα ήθελα να ζητήσω από τους συντονιστές μας να παρέμβουν έκαστος τρία λεπτά. Κύριος Κρισιάνης, εκ μέρους του ΕΛΚ. Κύριος Κάρινς. Ε, πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Βεβαίως δεν θέλω να σπαταλίσω το χρόνο μου να κάνω σχόλια, αλλά θέλω να σας κάνω ερωτήσεις. Αναφερθήκατε στην ουδετερότητα των δικτύων στο, στην περιαγωγή, ε, θέματα που μας απασχολούν όλους μας. Όσον αφορά την ουδετερότητα των δικτύων, θέλω να ρωτήσω το εξής. Εμείς ως ε, ευρωβουλευτές ε, βομβαρδιζόμαστε από διαφόρων ειδών συμφέροντα. Οι μεν λένε ότι πρέπει να ανοίξει ο κλάδος για τον καταναλωτή, από την άλλη όμως οι βιομηχανικοί κύκλοι λένε και εμείς πώς θα αποκομίσουμε χρήματα για να κάνουμε τις απαραίτητες επενδύσεις. Και γι' αυτό ερωτώ πώς μπορεί να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή ισορροπία έτσι ώστε από τη μια πράγματι να διατηρηθεί αυτό το άνοιγμα, από την άλλη όμως να συνεχίσει να υπάρχει και ενδιαφέρον εκ μέρους της βιομηχανίας για να προβαίνει σε απαραίτητες επενδύσεις. Σας είπα τρία λεπτά για τον κάθε συντονιστή, Ήταν πολύ πιο σύντομος και Γι' αυτό ε, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Επόμενος από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ο κύριος Νίκα. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, στη δική σας την παρέμβαση επισημάνατε ότι η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών βρίσκονται σε σκληρό ανταγωνισμό ανάμεσά τους ε, αλλά και απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει και αγορά του 4G και την προηγούμενη χρονιά η κυρία Νέλη Γκρός ε, ε, σε μια επιστολή αναφέρει ότι για το 4G στο 4G ανησυχεί μόνο το 6% της αγοράς. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι στον τομέα αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή, μόνο το 6% της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. Και ένας λόγος από τους σημαντικότερους λόγους που αναφέρθηκε για αυτή την αποτυχία στην Ευρώπη έχει σχέση με το γεγονός ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες έδρασαν ταχύτατα και ο άλλος λόγος ήταν ότι οι ρυθμιστικές αρχές κατέληξαν σε μια στάση που δεν ευνοεί την εξέλιξη σε αυτόν τον τομέα. Η τεχνολογία 4G, 4G δεν ενισχύθηκε, δεν στηρίχθηκε, κανείς δεν προώθησε αυτήν την τεχνολογία. Τώρα βέβαια γίνεται λόγος για νέες τεχνολογίες, για το 5G, 5G. Και θέλω λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Αν μέχρι τώρα είχαμε αποτυχία όσον αφορά τις ε, δραστηριότητες ε, των ρυθμιστικών αρχών, πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε στην επόμενη γενιά στο 5G και τελικά ε, το 4G, το 4G, πώς είναι δυνατόν να το βελτιώσουμε έτσι ώστε τουλάχιστον στο μέλλον να επιτύχουμε κάτι παραπάνω. Πρόεδρος, επόμενος ομιλητής, ο κύριος Τοσανόφσκι. κύριε Πρόεδρε. Συζητήσαμε τα έγγραφα τα οποία έχουν σχέση με την ε, διεύρυνση για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση σε διαδίκτυο, σε ίντερνετ υψηλής ταχύτητας. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε, κάποιος να μας πει τελικά Πώς θα πάει η Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα, σε αυτό το θέμα. Γιατί υπάρχουν πολλές διαφορές. Υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που τα καταφέρνουν καλύτερα, που είναι πολύ πιο προχωρημένες σε σχέση με άλλες, οι οποίες ε, δυστυχώς ε, απέτυχαν να διασφαλίσουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους υποδομές. Και εδώ δεν τίθεται τόσο θέμα των μεγάλων πόλων όσο των ε, μικρότερων της επαρχίας. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια σχετική έκθεση, ένα σχετικό απολογισμό. Πριν από τις εκλογές εγκρίναμε κάποιες αποφάσεις, αλλά θα θέλαμε να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για να γνωρίζουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξή μας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβασή μας στο διαδίκτυο. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής, Φρέντρικ Φέντερλεϊ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και για την εισήγηση που ακούσαμε. Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις πολύ σημαντικές ε, για την ομάδα μας, τους φιλελευθέρου. Μιλάμε για πάρα πολλά εκατομμύρια ανθρώπων που δεν προχωράνε στις επιχειρήσεις τους γιατί έχουμε διαφορετική νομοθεσία ε, στις διάφορες χώρες. Σε εμά ας πούμε στη Σουηδία είναι πολύ δύσκολο να απευθυνθούμε στο σύνολο της ε, ευρωπαϊκής αγοράς. Προχωρώντας την ψηφιακή εποχή βλέπουμε η δημοκρατία, οι υπηρεσίες υγείας, ε, τα φορολογικά, η πρόσβαση στα πανεπιστήμια, όλα αυτά έρχονται πιο κοντά στον πολίτη, στο βαθμό που έχει πρόσβαση ε, στο διαδίκτυο ή σε οπτικές σύνες. Στην Σουηδία πρέπει να σας πω έχουμε διαθέσει μεγάλα ποσά για να συνδέσουμε τις ε, μικρές πόλεις της επαρχίας με οπτικές ίνες στο μέλλον δεν θα μπορεί κανείς ε, να έχει πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες ε, εάν ε, δεν έχει διαδικτυακή σύνδεση. Σε κάποια νησιά που είναι δικά μας, έξω από τη Σουηδία, έχουμε σύνδεση 100% με οπτικές σύνες. Βεβαίως η Σουηδία είναι μια μεγάλη χώρα και εξακολουθούμε να έχουμε και εμείς αρκετές δυσκολίες. Εν πάση περιπτώσει, εάν το Κοινοβούλιο ή η Κομισιόν ε, δεν προωθήσουν την ε, κοινή αγορά, πάρα πολλές επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης και πολλές επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να συρρυκνωθούν γιατί θα είναι πολύ χρονοβόρες οι διαδικασίες εφαρμογής των ε, διατάξεων. Θα ήθελα λοιπόν να μας σχολιάσετε κατά την άποψή σας ποιο είναι το βασικό καθήκον αυτού του νέου κοινοβουλίου στον τομέα της ε, παροχής ε, υπηρεσιών σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκ μέρους της Γκουε, η κυρία Έρνστ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για όλα αυτά που ακούσαμε και έχω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση αφορά στον Μπέρεκ και στον τρόπο εργασίας του φορέα. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε πόσο διαφανές είναι όλο αυτό το μόρφωμα. Μιλήσατε για μια ομάδα εμπειρογνωμόνων. Αυτή ε, πώς ακριβώς, ποια είναι η σύνθεσή της και τι είδου διαφάνειας και έλεγχος υπάρχει. Ίσως μπορείτε να μας ενημερώσετε καλύτερα για τα θέματα εργασίας του φορέα Μπέρεκ. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι εσείς ε, αναφερθήκατε στην εναρμόνιση. Η εναρμόνιση ως στόχος και οι δυσκολίες που συμβαδίζουν με την εναρμόνιση. Και θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω το θέμα των ε, προσωπικών δεδομένων και της προστασίας τους. Τι ρόλο παίζει αυτό για σας, τι σκοπεύετε να κάνετε από αυτού. Και τρίτο θέμα που με ενδιαφέρει είναι η ουδετερότητα του διαδικτύου. Ε, και εδώ ε, είχαμε πάρα πολλές αντιπαραθέσεις, διαφωνίες, η ουδετερότητα του διαδικτύου δεν είναι δεδομένη. Και εσείς τι πιστεύετε, τι μπορούμε να κάνουμε για να την εξασφαλίσουμε. Αυτά τα τρία ερωτήματα παρακαλώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν βλέπω τον κύριο Τούρμες για να λάβει το λόγο εκ μέρου των ε, Πρασίνων. Ας πάμε λοιπόν ε, στην ε, Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Ο κύριος Ταμπουράνο παρακαλώ. Εγώ θα ε, αναφερθώ, θα λάβω το λόγο στην επόμενη συζήτηση που είναι περίπου παρεμφερής γιατί πρόκειται για το ψηφιακό θεματολόγιο. Κύριε εκπρόσωπε του Μπέρεκ, ακούσατε λοιπόν τον πρώτο γύρο ερωτήσεων και τώρα μπορείτε αν θέλετε να λάβετε το λόγο, να απαντήσετε. προσπαθήσω να απαντήσω σε ερωτήσεις που ήταν και πάρα πολύ εύστοχες, με εντυπωσίασαν οι ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν συντομότερο στις απαντήσεις μου. Σε ό,τι αφορά την ουδετερότητα του είπατε τι νομίζουμε και τι πράττουμε από αυτού. Να πω καταρχάς ότι ήδη το 2012 σε μια επίσημη γνωμοδότηση του Ομπέρεκ είπαμε ε, τι σκεφτόμαστε. Ε, είχαμε εκδώσει μια δήλωση που ε, ανέφερε πόσο σημαντικό είναι να είναι ανοιχτό το διαδίκτυο και να υπάρχει δυνατότητα επιλογής. Θέλουμε, ξέρετε τι γίνεται στη διασύνδεση μεταξύ ενός πομπού και ενός δέκτη. στο διαδίκτυο συνδέεται κάποιος και πληρώνει για την πρόσβαση και βέβαια έχει και ελεύθερη πρόσβαση σε ό,τι είναι ελεύθερο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό. Και έρχεται το εξής ερώτημα. Τα προβλήματα με την πρόσβαση πώς θα αντιμετωπίσουμε. Το πρώτο, σημαντικό είναι να υπάρχει διαφάνεια και ο τελικός χρήστης ε, να γνωρίζει τι αγοράζει και τι δεν αγοράζει. Η διαφάνεια λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική. Το επόμενο που λέγαμε στην γνωμοδότησή μας έχει να κάνει ε, με το ευρύτερο θέμα του ανταγωνισμού. Το έχουμε δει πολλές φορές στην Ευρώπη. Ακούμε ότι για το voice over IP θα υπάρξει περιορισμός ε, πρόσβασης και κάποιοι ανταγωνιστές ε, λένε εμείς δεν θα περιορίσουμε την πρόσβαση αν έχει επιλογή ο καταναλωτές, καταναλωτής, η εταιρεία λέει ότι θα περιορίσει την πρόσβαση, μετά όμως επειδή δεν θέλει να χάσει την πελατεία, ανοίγει ε, την πρόσβαση και πάλι. Επίσης, η νομοθεσία μας δίνει τη δυνατότητα να ορίσουμε τη διεθνή πρόσβαση αλλάζει και το διαδίκτυο, πρέπει να έχετε υπόψη και εμείς θα πρέπει να παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις. Να εξετάζουμε τα διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα. Γιατί είχαμε ένα πυλώνα αρχικά, όπου ο ίδιος χειριστής, ο ίδιος φορέας παρήχε όλες τις υπηρεσίες, ενώ τώρα έχουμε δύο πυλώνες και αλλάζουν συνεχώς τα πράγματα και η μορφή. Δεν μπορώ να σας πω αν σήμερα και σε πέντε χρόνια το διαδίκτυο θα είναι το ίδιο. Και είναι σημαντικό να δώσουμε δυνατότητες ε, να υπάρξουν και στο μέλλον εξελίξεις. Θέλουμε να δούμε λοιπόν και με την ομοθεσία τι μπορούμε να κάνουμε ως Μπέρεκ, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την τεχνολογία σε τρία-τέσσερα χρόνια, για το φάσμα. Αυτό το δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Μπέρεκ. Το επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη Σουηδία, για να δώσω ένα παράδειγμα, 90 ίσως και 100% των οικοκυριών έχουν 4G. Ε, και σε πολλές άλλες χώρες ε, έχει εισαχθεί. Οι παραδείγματος χάρη δεν είχαν ούτε 3G. Μέχρι στιγμής ε, δεν είναι ικανοποιητικέ οι λύσεις με το 3G και υπάρχουν κάποιες διαφορές. Σε ό,τι αφορά το φάσμα, θέλω να σας πω ότι το ψηφιακό μέρισμα είναι κάτι σημαντικό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν Επειδή κάποιος αναφέρθηκε σε κάποια γνωμοδότηση, σε κάποια αναφορά, πρέπει να σας πω ότι εμείς ως τεχνοκράτες κάνουμε πολλές αναφορές για τις χώρες ε, και η Κομισιόν κάνει πολύ καλή δουλειά, αναλύει, μελετά τις ε, μεμονωμένες χώρες και την κατάσταση που ισχύει. Πείτε μας τι θέλετε συγκεκριμένα και να έρθω και στην ερώτηση που μετέθη. Τι είναι το σημαντικότερο για το Κοινοβούλιο. Ε, με ικανοποιεί πολύ που τέθη αυτή η ερώτηση, αλλά πρέπει να σας πω ότι έχω μεγάλο σεβασμό για τους ερετούς άρχοντες. Εσείς είσαστε αυτοί λοιπόν που θα πρέπει να καθορίσετε το ρυθμό. Εγώ συμφωνώ με τη σημασία για τη δημοκρατία, για την ανάπτυξη, για την παιδεία. Οι αγροτικές περιοχές είναι μία πρόκληση πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος. Άρα, ίσω το σημαντικότερο δεν είναι να γίνει μια έρευνα πάνω σε αγροτικέ προχέ για να ξέρουμε ακριβώ τι γίνεται, αλλά να συνεχιστεί ο διάλογο. Αυτή θα ήταν η απάντηση. Τώρα, ο Μπέρικ προσπαθεί να είναι ένα διαφανή οργανισμό και νομίζω ότι είμαστε όλο και πιο διαφανεί. Τον Οκτώβριο θα έχουμε εδώ στις Βρυξέλλες μια συζήτηση μεταξύ των ε, ενδιαφερομένων 16 Οκτωβρίου. Είστε όλοι προσκεκλημένοι. Πολλοί θα συμμετέχουν και οι ομάδες ε, εμπειρογνωμόνων προετοιμάζονται. Είναι εκπρόσωποι των ε, εθνικών ρυθμιστικών αρχών αυτοί οι εμπειρογνώμονες. Και παραλαμβάνω ότι πάντοτε προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο διαφανείς. Επίσης αντιμετωπίζουμε τα πολύ σημαντικά ζητήματα της προσωπικής σφαίρας, της ε, παρακάτης κάποιων δεδομένων, της φύλαξης δεδομένων. Απόψεις έχουμε και εξετάζουμε όλα αυτά τα θέματα, αλλά δεν μπορούμε να επηρεάσουμε, δεν έχουμε αρμοδιότητα. Είμαι από το 2010 στον Μπέρεκ, ήμουν και ρυθμιστής, εθνικός ρυθμιστής ε, στη Σουηδία. Μας χτύπησε πριν από κάποια χρόνια η οικονομική κρίση, κάτι που σε πολύ σοβαρά προβλήματα σε πολλούς. Η εναρμόνιση, γιατί με ρωτήσατε, νομίζω ότι εξελίσσεται, βελτιώνεται αυτή η διαδικασία. Βλέπουμε ότι κάποιες χώρες χρησιμοποιούν ελαφρά διαφοροποιημένες μεθόδους. Η βάση είναι ίδια. Βέβαια δεν μας ικανοποιεί αυτό. Θέλουμε να υπάρξει βελτίωση γιατί έχουμε προκλήσεις και από την Ασία και από τη ΣΥΠΑ. Και το σημαντικότερο, όλοι θα πρέπει να έχουν την παγκόσμια πρόσβαση το συντομότερο δυνατό για να έχουν επιλογή. Νομίζω ότι απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις. Αν ξέχασα κάτι παρακαλώ να μου υπενθυμίσετε for your explanations and um, your remarks. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συζήτηση. Συνεχίζεται η συζήτηση, ευρωβουλευτές, από διάφορα ομάδες, ο κύριος Χόκμαρκ πρώτα. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την παρουσία. Τρεις ερωτήσεις έχω. Η πρώτη μου αναφέρθηκε και κάποιος νωρίτερα σε αυτήν έχει να κάνει ως εξής. Ε, μας προτείνατε να σας δώσουμε κάποιες ιδέες για εκθέσεις που θα κάνετε. Λοιπόν, αν κάνετε καλή δουλειά όσον αφορά την δετερότητα των δικτύων, την καλή ισορροπία. Δηλαδή, ναι, να είναι ανοιχτό το διαδίκτυο, αλλά να υπάρχουν και ειδικεύσει. Νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας για να πετύχουμε σαφήνεια στην νομοθεσία που προχωράει. Αυτό είναι το πρώτο, γιατί συγκρίσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική. Διστάζω πάντα, γιατί πάντα διαλέγουμε τα στατιστικά δεδομένα που μας δείχνουν καλύτερους και νιώθουμε ικανοποιημένοι από αυτό. Ή θέλουμε να αποδείξουμε το αντίθετο, ότι εμείς πάμε πίσω και όλοι οι άλλοι είναι καλύτεροι. Οπότε ανάλογα διαδεύουμε στατιστικά δεδομένα. Γι' αυτό λοιπόν για μένα είναι πιο σημαντικό να εντοπίσουμε τις αδυναμίες μας. Γιατί είμαστε σε έναν αγώνα με κινούμενους στόχους. Δεν ξέρουμε πώς θα έχει η κατάσταση σε πέντε χρόνια πράγματι. Αλλά πρέπει να βασιστούμε σε αυτά που ξέρουμε, στην ποιότητα, την ποσότητα, κλπ. κλπ. Θα ήταν λοιπόν καλό αν ο οργανισμός Μπέρεκ μπορούσε να έχει μια ισορροπημένη έκθεση που να αναφέρει τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Τρίτον, όσον αφορά τον ίδιο τον Μπέρεκ. Από την εμπειρία σας, τα τελευταία χρόνια, στις δραστηριότητες του οργανισμού, τι νομίζετε ότι θα έπρεπε να αλλάξει ώστε ο Μπέρεκ να μπορέσει να λειτουργήσει πλήρως και να φέρει σε πέρας πλήρως το ρόλο του που είναι ένα ευρωπαίο Ευρωπαίος ρυθμιστής. Τι θα θέλατε να αλλάξει για να έχει ο οργανισμός καλύτερες, περισσότερες πιθανότητες να φέρει σε πέρας τις αλλαγές που χρειαζόμαστε στην ψηφιακή αγορά. Ευχαριστούμε κυρία Τόγια τώρα. Κοιτάξτε, η δική μου ερώτηση έχει σχέση με το τελευταίο σκέλος της ε, παρέμβασης του συναδέλφου. Και ε, θέλω να ρωτήσω κάτι οι δραστηριότητες ε, του Μπέρεκ. Εμείς ανέκαθεν τη στηρίζαμε αυτή ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θεωρούμε ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ε, όσον αφορά γενικά τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς σε αυτόν τον τομέα. Και θέλω να ρωτήσω, γιατί και εσείς το είπατε, το, ο Μπέρεκ για να αναπτύσσει καλύτερα τις δραστηριότητές του. Τι θα ήταν πιο χρήσιμο να λάβει η χώρα, τόσο στις σχέσεις του με, τις, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και με τις εθνικές ε, ρυθμιστικές αρχές. Εντάξει, δεν είσαστε εσείς ο νομοθέτης, αλλά θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι είναι εκείνο που θα μπορούσε να βελτιωθεί, να βελτιωθεί στις σχέσεις με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά σας παρακαλώ πολύ να μου απαντήσετε επί όχι μια ξύλινη τυπική απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ξέρετε ότι ο κόσμος είναι άνισος και το διαδίκτυο αποτελεί μέρος του κόσμου, οπότε και το διαδίκτυο δεν ε, προσφέρει ισότητα. Όσον αφορά την ανωνυμότητα στο διαδίκτυο, εγώ θέλω να ρωτήσω. Οι πολίτες, όπως δουλεύουν με το διαδίκτυο, είτε αγοράζουν, είτε στέλνουν μηνύματα, ελέγχονται συνεχώς. Τους παρακολουθεί το διαδίκτυο και τα δεδομένα αυτά διατηρούνται από τις κυβερνήσεις, από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Θέλω λοιπόν να ξέρω ποια είναι η θέση του Μπέρεκ, αν έχει κάποια θέση όσον αφορά το θέμα της ανωνυμίας και κατά πόσο θεωρεί ή όχι ότι θα έπρεπε να αναλάβουμε κάποια δράση για να προστατεύσουμε τον ιδιωτικό βίο και την ανωνυμία των Ευρωπαίων πολιτών σε αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστούμε. Τεντίτσκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αναφερθήκατε στην νομοθεσία όσον αφορά την ουδετερότητα των δικτύων και την περιαγωγή. Φυσικά και αντιλαμβάνομαι και έχω κάθε σεβασμό για τη θέση σας, που είναι η επίσημη θέση. Είσαστε όμως ένα σώμα ανεξάρτητων ρυθμιστών, σωστά. Οπότε γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν με το Συμβούλιο όσον αφορά την νομοθεσία και θα αρχίσουμε να έχουμε και συνεδριάσεις τριμερούς διαλόγου. Τα δικά σας τα μέλη, τι εντοπίζουν ως δυσκολία, ποιες δυσκολίες ανοιχνεύουν ότι θα εμφανιστούν από πλευράς του Συμβουλίου, τι ακούγεται δηλαδή όσον αφορά τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε στις συνονίσεις αυτές με το Συμβούλιο. Ευχαριστούμε. Γκρίφιν, η κυρία Γκρίφιν. Ευχαριστώ πολύ. Αναφερθήκατε σε μεγάλη ταχύτητα ευρυζωνικότητας για όλους. Εσείς πώς αξιολογείτε την επιτυχία όσον αφορά τους ποιοτικού δείκτες και όχι μόνο βάσει του κόστους να έχουν όλοι, να έχουν και τα άτομα με αναπηρίες, άτομα στο περιθώριο. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Μπαγιώνη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την παρουσίαση, λέει ο κύριος Μπόνη. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, συμφωνώ απόλυτα για το ότι πρέπει να επανέλθουμε στη συζήτηση όσον αφορά την ουδετερότητα των δικτύων και να προσπαθούμε να πετύχουμε κάποια ισορροπία ανάμεσα στις προσδοκίες των ε, πολιτών, των φορέων, ε, των χρηστών. Να ξέρουμε τι γίνεται από πλευράς τεχνολογίας, τι γίνεται από πλευράς ε, λειτουργίας. Τι λέτε για αυτή τη δυνατότητα. Δεύτερη ερώτηση. Έχει να κάνει με αυτό που είπατε, ότι χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα όσον αφορά τον ανταγωνισμό της Ευρώπης σε σχέση με άλλα σημεία του κόσμου. Συμφωνώ βέβαια, απολύτως, αλλά πρέπει να είμαστε πιο θαραλέοι όταν μιλάμε για ρυθμίσεις. Αν θέλουμε παγίωση και θέλουμε ρύθμιση, τι θέλουμε, θέλουμε ευρωπαϊκή ρύθμιση Χωρίς σύνορα. σε ευχαριστούμε. Δεν βλέπω κανέναν άλλον να ζητάει το λόγο. Οπότε, παρακαλώ. Κάνετε εύκολη τη ζωή μου, ξέρετε. Θα αρχίσω με το εξή. Υπάρχει ένα όριο, μια διαφορά ανάμεσα στη δικιά σας τη δουλειά και τη δικιά μου τη δουλειά. Εγώ είμαι ταπεινός σας υπηρέτης. Βοηθώ για την νομοθεσία. Οι γραφειοκράτες που προσπαθούμε να την κάνουμε όσο γίνεται καλύτερη την νομοθεσία αυτή, βασισμένη όμως στις δικές σας αποφάσεις. Εσείς κάνετε τις πολιτικές συζητήσεις. Και εμείς τις εφαρμόζουμε, γι' αυτό φτιάξατε τον Μπέρεκ. Τώρα, αναφερθήκατε στις στατιστικές. Εγώ μίλησα για αυτές γιατί ξέρω ότι φέτος θα ακούσετε πολλά για συγκρίσεις και πρέπει κανείς να ξέρει ότι γίνονται πολλές συζητήσεις και όντως μπορεί κανείς να συγκρίνει πράγματα με διαφορετικούς τρόπους. Οπότε συμφωνώ ότι υπάρχουν ε, διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Πράγματι και αυτό πρέπει να το διορθώσουμε. Νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι η αγορά αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό. Όταν πάμε στο 4G, πολύ σημαντική αλλαγή αυτή για τους πολίτες, ε, βλέπουμε ότι εδώ παραβαίνει και το φάσμα. Και αυτό γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Άρα πρέπει να γίνουν τέτοιες συζητήσεις και αυτά που συζητάμε για το θέμα του ιδιωτικού βίου ε, και τα λοιπά δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα. Στις συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολλές φορές λέμε πώς ε, θα συναρμολογήσουμε το πακέτο αυτό. Υπάρχουν πολλά πράγματα που εμεί δεν κάνουμε καθόλου, όπως το IPR. Ποιος δηλαδή ελέγχει τα θέματα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Πώς θα είναι η αγορά σε μερικά χρόνια δεν το ξέρουμε. Το 2012 βγάλαμε κάτι που το ονομάσαμε Mid-Term Strategy. Μεσοπρόθεσμη στρατηγική και σε λίγους μήνες από πλευρά της Μπέρεκ θα πούμε τι πιστεύουμε ότι θα συμβεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια στην αγορά αυτή. Κάνουμε έρευνες και προσπαθούμε όντως να αντιληφθούμε πώς θα είναι η αγορά σε λίγα χρόνια. Έρχομαι τώρα στην ε, ουδετερότητα των δικτύων. Το βασικό στοιχείο της συζήτησης αυτής είναι ότι δεν ξέρουμε πώς θα είναι σε λίγα χρόνια. Στη Σουηδία έχουμε ετοιμάσει ένα νέο φόρουμ για την ουδετερότητα των δικτύων και καλούμε διάφορους ε, παράγοντες, φορείς από τη βιομηχανία, ειδικού, αλλά και καταναλωτές για να προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε ποιες θα είναι οι ανάγκες όλων των πλευρών. Και βάσει αυτού θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Τώρα, αυτό που μου άρεσε πολύ είναι που ρωτήσατε πώς μπορούμε να υπολογίσουμε την επιτυχία. Μα εξαρτάται από το στόχο που θέτουμε. Αν βάλουμε έναν εύκολο στόχο, όλοι τον πετυχαίνουμε. Το θέμα είναι ότι εσείς μας βάζετε στόχους σημαντικούς και εμείς είμαστε στον αγώνα να τους πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Πολλές συζητήσεις έχουν να γίνουν για την επιτυχία. Τη μετράμε μαζί σας, με τους πολίτες. Εγώ δεν έχω αντίρρηση να θέτετε υψηλούς στόχους για μας, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που θα σας πω αν έχουμε πετύχει όχι. Υπάρχει και ένα σχόλιο όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν συμφωνούμε πάντα μεταξύ μας, γιατί είμαστε ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Όταν λοιπόν κάποιος μας ρωτάει τη γνώμη μας, τι λέμε, τη γνώμη μας ως έχει. Αυτή η ανεξαρτησία που έχουμε είναι πολύ σημαντική και νομίζω ότι όλοι σέβονται την ανεξαρτησία αυτή του Μπέρεκ. Είτε συμφωνεί η Επιτροπή, είτε δεν συμφωνεί. Μερικές φορές διαφωνούμε και μαζί σας. Γι' αυτό και είναι ωραίο πράγμα να είναι κανείς ρυθμιστής. Είναι με πολλές εντάσεις δουλειά αυτή. Πάντως, έχουμε πολύ καλές σχέσεις εργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμείς στον ΠΕΡΕΚ. Ναι, μερικές φορές μπορεί να διαφωνούμε μαζί τους. Αλλά αυτή τη δομή επιθυμήσατε εσείς. Να γίνονται συζητήσεις για τον καλύτερο τρόπο που έχουμε για να προχωρήσουμε. Όντως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε πάρα πολλές συζητήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξάλλου είναι παρατηρητής, παρίστατος παρατηρητής της δικές μας συνεδρίες. Τώρα, η αγορά ηλεκτρισμού, για παράδειγμα, είναι όπως οι τηλεπικοινωνίες. Μιλάμε για την πρόσβαση σε ένα σπίτι. αν δεν μπορώ να διαλέξω προμηθευτή, δεν έχει νόημα, πρέπει να μπορώ. Και η μεγαλύτερη αλλαγή εδώ είναι ότι έχουμε βγει από την λογική του μονοπωλίου σε μια άλλη λογική, σε έναν άλλο κόσμο όπου υπάρχει υποδομή από τη μια μεριά και κάποιος άλλος προσφέρει τις υπηρεσίες. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε γιατί μπορεί να καταλήξουμε να έχουμε στις υποδομές πολύ καλό ανταγωνισμό, αλλά μονοπόλια όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών. Υπάρχουν πολλές μεγάλες εταιρείες που έχουν μεγάλο τμήμα της αγοράς στο διαδίκτυο σήμερα. Γι' αυτό τις συζητήσεις αυτές και τις μερικές δεν πρέπει να τις κάνουμε πριν προχωρήσουμε και πούμε ότι μία πλευρά είναι πιο σημαντική από την άλλη, υποδομές δηλαδή οι υπηρεσίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες ε, τις ε, εξηγήσεις, τις παρατηρήσεις, την παρουσία σας εδώ στο Κοινοβούλιο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η συνεργασία μεταξύ του Μπέρεκ και προσωπικά μεταξύ ημών και ημών διασφαλίζει και την καλή συνεργασία μεταξύ των αριθμιστικών αρχών των κρατών μελών. Ελπίζουμε η εξαιρετική συνεργασία να συνεχιστεί γιατί αυτό θα διευκολύνει πάρα πολύ τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Uh, λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο σημείο 6 της Μερισιάς Διάταξης ή το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, την παρουσίαση του Γενικού Διευθυντή Ρομπέρ Μαντλά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. So, well, uh, uh digit, Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη λοιπόν. Στόχος είναι να επανεκκινήσει η ευρωπαϊκή οικονομία, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να εκμεταλλευτούν τι ψηφιακές τεχνολογίες. Έχουμε 7 εμβληματικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της ε, Ευρώπης 2020 της στρατηγικής αυτής που στόχο είχε μια ευφυή ανάπτυξη για όλους. Το ψηφιακό θεματολόγιο το διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση για τα δίκτυα της τηλεπικοινωνίας Κομισιόν. Θέλω να καλωσορίζω τον κύριο Ρομπέρ Μαντλά, τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔ Connect. Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που ξαναέρχομαι στην ανασυγκροτηθήσα επιτροπή σας, γιατί δεν υπάρχουν μόνο νέο εισερχόμενοι, υπάρχουν και πάλι γνώριμοι. Θέλω να σας συγχαρώ και εσάς που ε, εκλεκτικά του Πρόεδρου. Είμαστε 1100 υπάλληλοι στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο Θεωρούμε ότι αυτή η Επιτροπή είναι από τις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, που είναι και στο επίκεντρο των δικών μας δράσεων. Θεωρούμε ότι αν η καινοτομία ε, ξεκινά από την Ευρώπη με τη χάραξη ευρωπαϊκών πολιτικών στρατηγικών και με τον προϋπολογισμό, αν είναι η κοινωνία έτοιμη για την καινοτομία, μπορούμε να πετύχουμε και εμείς ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και η ψηφιακή τεχνολογία το ψηφιακό τεματολόγιο είναι ένα σημαντικό κομμάτι της προσπάθειας για καινοτομία και έρευνα. Θα ξεκινήσω με την ομαλή μετάβαση. Είμαστε υπάλληλοι οι οποίοι προσπαθούμε και με τη δική σας βοήθεια γιατί θα έχουμε τη μετάβαση τον Νοέμβριο από την Κομισιόν Μπαρόζο 2 στην Κομισιόν Juncker 1 πρέπει να συνεργαστούμε και έχουμε και μια πολύ βεβαρημένη μερίσια διάταξη. Θα έχουμε την εκδήλωση για τη ε, ψηφιακή τεχνολογία. Θα ακούσετε τον Γενικό Διευθυντή της ΕΝΙΖΑ. Δεκαετία πλέον κλείνει αυτός ο οργανισμός τον Οκτώβριο. 11 και 17 επί, 17 έχουμε πολλά, πολλά την επόμενη, τις επόμενες εβδομάδες που φαντάζομαι θα σας ενδιαφέρουν. Έχω αφήσει στην γραμματεία ένα τετρασέλιδο έντυπο που αναφέρει τις ημερομηνίε και τις εκδηλώσεις. Όποιος θέλει μπορεί να το μελετήσει. Δεν περιμένουμε λοιπόν. Ήδη από τώρα δραστηριοποιούμε. Θα ξεκινώ λοιπόν πρώτα απ' όλα με τις ευρυζωνικές υποδομές και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Ο προλαλής σας ε, από τον Μπέρεκ μίλησε ε, γι' αυτό και την εβδομάδα αυτή θα έρθουν και κάποιοι εμπειρογνώμονε από τη δική μα Γενική Διεύθυνση. Να ξεκινήσω με τι υποδομέ. Το όραμα τη σημερινή Επιτροπής ήταν να δώσει στην Ένωση όλες τις υποδομές για να μπορέσει να ανθίσει, για να έχουμε ε, αξιοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Και να μην έχουμε υποδομές μόνο σε πλούσιες ε, πόλεις και αστικά κέντρα, αλλά σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουμε να κλείσουμε τα χρηματοδοτικά κενά που υπάρχουν ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του προηγούμενου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας. Υπάρχουν μεγάλα κενά, τεράστια κενά. Και το χάσμα αυτό, ένα ευρώ στα πέντε έχει ε, μειωθεί. Το 80% του χρηματοδοτικού κενού για την επίτευξη των στόχων μας σε ό,τι αφορά την ευρυζωνικότητα δεν έχει επιτευχθεί ακόμη, το 80%. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να έχουμε υπόψη. Δεν μιλάμε μόνο για δημόσια κονδύλια, μπορεί να πρόκειται για νέους χρηματοδοτικούς ε, οργανισμούς. Θέλουμε να έχουμε και ένα καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να εντάξουμε και τις ιδιωτικέ επενδύσεις, αλλά δεν υπάρχει επαρκή ισορροή ε, ώστε να έχουμε τις επενδύσεις που τόσο χρειαζόμαστε. Στις ε, δαπάνες λοιπόν για τις ευεζονικές υποδομές και έχουν και τον κανονισμό για την ενιαία αγορά. Είναι ένα κομμάτι σε αυτό τον κανονισμό που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Δεύτερον, τι κάνουμε με την ευεζονικότητα ανταλλάσσουμε όχι μόνο εικόνες ε, και βίντεο από γατάκια, αλλά θέλουμε να κάνουμε πιο αποτελεσματικές, υγιείς, ασφαλείς της πόλεις μας, τα σχολεία μας ε, και όλα τα εκτίρια. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο ταχείς, πιο γρήγοροι. Αυτό είναι ένα μήνυμα της, του ψηφιακού θεματολογίου και νομίζω ότι ο πρόεδρος Γιούνκερ το έχει πει. Δεν είναι όλα διασυνερικά ούτε όλα ευρυζωνικά. Έχουμε και, ε, παραδείγματο χάρη, τις τιμές ε, στο ταχυδρομείο. Τα τέλη, τα ταχυδρομικά διαφέρουν. Οι αδερφοί μου δεν πληρώνουν τα ίδια με τον αδερφό μου που ζει σε διαφορετικό μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι σημαντικά λοιπόν αυτά και για το ηλεκτρονικό εμπόριο και για την ευρυζωνικότητα. Αλλά και όλοι μας ε, όταν ψωνίζουμε. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε έναν ευφύ διχρηματοδοτικό μηχανισμό. Έχουμε πρόοδο επιτελέσει τα τελευταία χρόνια, αλλά πρέπει να επιτελέσουμε ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο. Το τρίτο που θέλω να αναφέρω είναι η έρευνα, που είναι ένας κοινό στόχος. ορίζοντας 2020 νομίζω ότι είναι πιο ρηξικέλευθο πρόγραμμα από αυτό που έχει καταλάβει ο κόσμος. Θα πρέπει να αναλάβει βέβαια πιο υπεύθυνη έρευνα, να είναι πιο εύκολο να το χρησιμοποιούσουν οι ερευνητές, οι ΜΜΕ, ε, ερευνητικοί φορείς. Πρόοδο έχουμε επιτελέσει, αλλά δεν έχουμε ακόμη επιτύχει το στόχο μας εντελώς. Υπάρχει ένα πρόβλημα να έχουμε ελλείψεις οικονομικές, να μην επαρκεί ο προπολογισμό. Το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε προβλήματα ε, το γύρο το 2014. Όταν θα λάβουμε αποφάσεις λοιπόν για το 2015, ε, πρέπει να βλέπουμε ότι το, το πρόβλημα ήδη υπάρχει. Αν δεν μπορούν να πληρωθούν τα τιμολόγια, δεν θα είναι και ε, αυτό ένα καλό κίνητρο για τους ερευνητές. Η ψηφιακή έρευνα για την καινοτομία επίσης πηγαίνει πολύ καλά η επανεκβιομηχάνηση μέσω της καινοτομίας στο ψηφιακό κόσμο είτε για τους μια ημιαγούς τελευταίας γενιάς είτε για το ε, υπολογιστικό νέφος είτε για άλλους τομείς. και για την κυβερνοασφάλεια εκβιομηχάνηση μπορούμε να τα καταφέρουμε πολύ καλύτερα σε αυτούς τους τομείς. Θα Ήθελα λοιπόν να περιουσώ σε αυτή τη σύντομη παρουσίαση, γιατί νομίζω ότι σημαντικό είναι να βάλουμε κάποιους τίτλους και να εμβαθύνουμε στη συνέχεια εκεί που οι βουλευτές θέλουν να θέσουν ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Uh, thank you. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Διευθυντά. Θα δώσω το λόγο στους συντονιστές. Ο κύριος Κριστιανής Κάρινς από το Έλκυνο Πρώτος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για την εισήγησή σας. Ε, χαρήκαμε πάρα πολύ που ήταν ε, σύντομη. Αυτό δεν συνηθίζεται. Τώρα, μία ερώτηση για την ψηφιακή κοινή αγορά. Με βάση τα στοιχεία που μας παρουσιάσατε, το 7% επιτυγχάνει περίπου το στόχο 12% είναι το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, είναι κάτω από το ίμιση του στόχου. Και θέλω να ρωτήσω ποιος είναι, ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο που υπάρχει σε όλα αυτά και τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ε, να συγκεντρώσουμε κάποιες ερωτήσεις και μετά αν θέλετε μπορείτε να απαντήσετε. Νταν Νίκα εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών παρακαλώ. Κύριε Γενική Διευθύντα, έχω μια ερώτηση σχετικά με τα 4G και επίσης ε, θέλω να ρωτήσω πώς μπορούμε να διαδώσουμε το διαδίκτυο στο σύνολο της υπέτρου. Αν κατάλαβα όμως καλά, η Ευρώπη δεν είναι αρμόδια για όλα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι δεν είναι αρμόδια γι' αυτό, αλλά ούτε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και διερωτώ με κατά πόσο αυτή την ερώτηση μπορούμε να τη θέσουμε στο Συμβούλιο. Ποιος είναι τελικά αρμόδιος. Πάντως ε, αυτό το θέμα έχει σχέση με το ψηφιακό θεματολόγιο. Ε, γιατί ε, χωρίς ευρυζωνικότητα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ψηφιακό θεματολόγιο σε καμία χώρα της Ευρώπης. Και θέλω να ρωτήσω κάτι για τα κονδύλια. Γιατί πολλά από τα κονδύλια που διατίθενται τα διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων. Και ερωτώ, ποιο είναι το ύψος των κονδυλίων που προβλέπετε από εσάς και μήπως αξίζει το κόπο να επενδυθούν περισσότερα χρήματα. Και γι' αυτό λοιπόν σχετικά με το 4G, ε, το 4G, Θέλω να γνωρίζω κατά πόσο αυτό το θεωρείτε ως βάση του ψηφιακού θεματολογίου ή όχι. Μερικοί λένε ότι το κινητό 4G δεν είναι κινητό. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω προφανώς και έχει σχέση με τον ορισμό και διερωτώ με ε, κατά πόσον υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και τελική ερώτηση. Πιστεύετε ότι στη Γενική Διεύθυνση ε, για την Αγροτική Ανάπτυξη κάτι πρέπει να γίνει έτσι ώστε να λαμβάνονται διαφορετικές αποφάσεις και να επιτυγχάνουμε το στόχο μας με καλύτερο τρόπο. Πρόεδρος, ο κ. Τοσανόφσκι παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την εισήγηση που μόλις ακούσαμε μετά τις ε, διακοπές. Αυτή είναι η πρώτη συζήτηση που ακούμε για το ψηφιακό θεματολόγιο. Το ψηφιακό θεματολόγιο το εγκρίναμε στις αρχές του καλοκαιριού, περισσότερο κατά το τέλος της άνοιξης. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι δεν μπορούμε ήδη τώρα να έχουμε τα προσδοκούμενα αποτελέσματα. Όλα αυτά αφορούν και το πρόγραμμα ε, Horizon και ε, Connect. Παρότι λοιπόν περιορίσαμε τα κονδύλια, παρόλα αυτά ε, υπάρχουν κονδύλια τα οποία διατέθηκαν. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω πότε προβλέπετε ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πότε θα μπορούμε να δούμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και να γνωρίζουμε κατά πόσον επιτεύχθηκαν οι στόχοι μας ε, κυρίως σε σχέση με την ουδετερότητα του διαδικτύου. Και επίσης και με την ταχύτητά του ε, θα πρέπει να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Εσείς πότε το βλέπετε, για πότε το βλέπετε να έχουμε ε, μια άποψη, ένα συμπέρασμα ε, κατά πόσον επιτύχαμε ή όχι. Υπάρχει, ε, όπως σας είπα, το πρόγραμμα Connecting Europe μεταξύ άλλων και ενδεχομένως θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το πώς ε, εκταμιεύουν τα κονδύλια. Μήπως θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την κατανομή τους και πότε πιστεύετε ότι θα πρέπει να έχουμε μία σε βάθος συζήτηση ε, σχετικά με όλα αυτά τα θέματα. Εμείς την είχαμε προβλέψει τη συζήτηση για τις αρχές του έτους. Νομίζω όμως ε, ότι θα πρέπει να έχουμε μια διαφορετική ημερομηνία. Πρόεδρε και κύριε Γενικέ Διευθυντά, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς ε, και την Αντιπρόεδρο για την πολύ καλή δουλειά που κάνετε για να ε, προαχθεί το ψηφιακό ε, θεματολόγιο. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια πανευρωπαϊκή υποδομή και να εφαρμόζονται ευρωπαϊκά προγράμματα με ασφάλεια. Πρέπει να σας πω ότι εμένα με απασχολεί το γεγονός ότι παρότι μπορούμε να αγοράζουμε ε, και να χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικά τα αεροπορικά μας εισιτήρια. Παρόλα αυτά είμαστε υποχρεωμένοι να τα εκτυπώνουμε και να τα υπογράφουμε κιόλας εφόσον καλούμεθα να τα υποβάλουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί να μην είναι δυνατόν να ε, χρησιμοποιούμε τα ηλεκτρονικά έγγραφα και την ηλεκτρονική υπογραφή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό μπορεί να σας φαίνεται λεπτομέρεια, δεν είναι όμως, γιατί δείχνει ότι πρέπει να δουλέψουμε για να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σιλικιώτης, παρακαλώ. Όχι, η κυρία Έρνστ. Η κυρία Έρνστ εκ μέρους της ε, Γκουε. Όχι ως ε, συντονίστρια, αλλά αρμόδια ε, αν θέλετε για αυτό το θέμα. Υπάρχουν δύο θέματα τα οποία με απασχολούν. Βεβαίως, καταρχήν, αυτά όλα που μας είπατε ε, κατέστησαν ε, σαφή ότι μάλλον ε, βρισκόμαστε εδώ μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και σε οικονομικό και σε δημοκρατικό επίπεδο, αν θέλουμε να εφαρμόσουμε το ψηφιακό θεματολόγιο. Και βεβαίως όλα αυτά σε τελική ανάλυση συρρυκνώνονται στο οικονομικό και σε εμά υπάρχουν πάρα πολλά ελλείμματα στην ευρυζωνικότητα. Η ευρυζωνικότητα είναι καθοριστική σημασία. Και τίθε το εξή ερώτημα. Εσεί μιλήσατε για οικονομική φύσεω πρόβλημα και το ξέρουμε αυτό. Πράγματι είναι περιορισμένα τα οικονομικά και αυτά έχουν επιπτώσεις και αν δει κανεί ε, λιγάκι το μέλλον, εσείς πού ακριβώς εντοπίζετε τα προβλήματα λόγω του ότι δεν θα υπάρχουν ε, επαρκή κονδύλια. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Και το δεύτερο είναι, μάλλον και στη συνέχεια του πρώτου, είναι τι θα προκύψει από την έλλειψη οικονομικής υποστήριξης. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι επειδή υπάρχουν ε, οι κυβερνοεπιθέσεις, το κυβερνοέγκλημα, ε, προκύπτουν κάθε χρόνο τεράστιες δαπάνες. Μιλάμε για δισεκατομμύρια τα οποία χάνονται και θα ήθελα να ρωτήσω το εξή, η ασφάλεια του διαδικτύου. Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο για να έχουμε και καλύτερη προστασία από το κυβερνό έγκλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι πράσινοι τώρα δεν εκπροσωπούνται από ό,τι βλέπω. Ο κύριος Ταμπουράνου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πόσα λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας οι συντονιστέ. τρία λεπτά. Αν παρότι η τρια λεπτα αν παροτι υπάρχει ε, αύξηση στον τομέα αυτό κατά 12 περίπου Αυτό δεν ισχύει σε όλες τις χώρες, ε, ας πούμε στην Ιταλία. Και υπάρχουν δυστυχώς ακόμα ολιγοπόλια. Ε, οι περισσότερες συνδέσεις είναι ασύμετρες, η ταχύτητα του download είναι περιορισμένη και γι' αυτό δεν μπορούμε να έχουμε ικανοποιητικές υπηρεσίες αυτό που ενδιαφέρει είναι να έχουμε μια πραγματική ψηφιακή δημοκρατία χωρίς να επηρεάζει τα δικαιώματα των χρηστών. Πρέπει λοιπόν να ε, προτείνουμε κάποιες προσεγγίσεις bottom-up, ε, να αναλάβουμε κοινωνικές πρωτοβουλίες και αυτές να είναι πολύ πιο σημαντικές από τις τεχνολογικές. Εδώ αναφέρομαι ε, στο διαδίκτυο υπάρχουν οι τεχνολογίες peer-to-peer peer to peer και αυτά έχουν άμεση σχέση με τους ε, χρήστες. Οι χρήστες ε, προφανώς και εξαρτώνται από τα ελιγοπόλια και από την ε, ευρυζωνικότητα που διατίθεται από το κράτος. Παράδειγμα, στη δική μου, την, το σπίτι μου στη Ρώμη, μπορώ να έχω 23 MB ανά δευτερόλεπτο σε χαμηλή τιμή, σε μία, με μία όμως ταχύτητα που δεν είναι εγγυημένη και εν τόσο, είναι πολύ καλύτερη από άλλες περιοχές. Στην Πόντζα, σε ένα μικρό νησί της Ιταλίας, εκεί η ευρυζωνικότητα είναι διαδεδομένη και ίσως είναι και καλύτερη και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω μπορεί να υπάρχει κάποια ισορροπία όσον αφορά την ευρυζωνικότητα με χαμηλό κόστος αυτή να προσφέρεται και στην επαρχία που δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Was absolutely enough time, as you see. now we'll be... Ευχαριστούμε. Ωραία. Τώρα να ακούμε τις παρατηρήσεις σας μετά το δεύτερο αυτό γύρο. Ευχαριστώ πολύ. Ίσως δεν θα απαντήσω με τη σειρά. Θα προσπαθήσω όμως να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις και θα ξεκινήσω από το τέλος, από τον κύριο Ταμπουράνου. Από το 2010 μιλάμε για το πώς όλοι πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά δίκτυα. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έλεγα ότι είμαστε αυτοί που λιγότερο γνωρίζουμε. Περνώντας από διάφορες χώρες, έχω διαπιστώσει ότι οι λύσεις που έχουν διάφορες χώρες είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα για το πώς φροντίζουμε όλοι οι πολίτες να συμμετέχουν. Όλες οι χώρες το κάνουν, όλες οι χώρες το προσπαθούν. Προσπαθούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τους εθνικούς πρωταθλητές, τις καλύτερες λύσεις δηλαδή, και να προωθήσουμε αυτές τις εθνικές λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι κανένα μυστικό η Αντιπρόεδρος Κρούς είναι υπέρ αυτής της μεθόδου, δεν το κρύβω. Αλλά λέμε στις ε, διάφορες χώρες αυτή είναι η καλύτερη λύση, προσπαθήστε να την ε, εφαρμόσετε, αλλά μέχρι εκεί δεν μπορούμε να επιβάλλουμε με νομοθεσία δραστηριότητες από πάνω προς τα κάτω. Αυτό που με τη δικιά σας τη βοήθεια όμως έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε συζητήσει να σκιαγραφηθούν τα διάφορα στοιχεία της σημερινής κατάστασης και έτσι να καλύψουμε το ψηφιακό χάσμα. Αν όλοι θέλουν ευρωζενικότητα και τη ζητάνε τοπικά, τότε θα ξέρουμε πολύ καλύτερα ποιο θα είναι το κόστος. Έχουμε τώρα και σε αυτό που ρώτησε ο κύριος Νίκα. Δηλαδή, αν τα χρήματα υπάρχουν από τα διαφορετικά ταμεία, γιατί δεν μπαίνουν σε αυτό το τομέα. Από την αρχή του σχεδίου ανάκαμψης, οι επιδόσεις μας είναι χαμηλές όσον αφορά τη χρηματοδότηση σε τοπικό επίπεδο. Πρώτα απ' όλα προσπαθούμε ε, κάποια χρήματα από την Ήπεθρο να πάνε στην ευρυζωνικότητα, αποτύχαμε. Οι τοπικές αρχές που ξέραν πώς να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα ανάπτυξης της υπαίθρου, δεν μπόρεσαν να, να τα χρησιμοποιήσουν στην ευρυζωνικότητα και γύρισαν πίσω. Έτσι κι αλλιώς πάντως οι τεχνολογίες, οι τεχνολογίες είναι μια προτεραιότητα πάντα. 4-5% στην τελευταία χρηματοδοτική περίοδο ε, ήταν για τις ε, τεχνολογίες πληροφορικής, τώρα θα είναι 10% στην επόμενη περίοδο. Ξέρετε, μερικέ φορέ οι δρόμοι και οι γέφυρε, και δεν έχω τίποτα εναντίον δρόμων και γέφυρων, είναι κάτι πιο ελκυστικό από το ψηφιακό χάσμα. Ίσως γιατί είναι κάτι που μπορούν να δουν και να πιάσουν. Πάντως είναι θέμα λεγής νοοτροπίας. Η επόμενη πρωτοβουλία που θέλουμε να πάρουμε είναι να δουλέψουμε και σε τοπικό επίπεδο με τους διαφορούς φορείς, όχι μόνο δηλαδή εδώ με το Ευρωκοινοβούλιο, την ε, Περιφερειακή Επιτροπή, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Έτσι και ο κύριος Τεζονόφσκη το είπε αυτό. Έτσι ερχόμαστε στο θέμα των υποδομών και τον ε, κύριο Γιούνκερ, πώς το βλέπει, τα 300 εκατομμύρια που είπε. Και παρά τα χαμηλά ποσά που πηγαίνουν στην ευρωζενικότητα, ελπίζουμε ότι το όλο θέμα θα αποκτήσει μεγαλύτερη ε, σημασία. Ναι, το ψηφιακό χάσμα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει σε τοπικό επίπεδο να ενθαρρύνουμε τις τοπικές αρχές να ενισχύσουν την ευρυζωνικότητα. Έρχομαι τώρα και στο θέμα της ασφάλειας και ο κύριος Δοσνόφσκι και η κύριε Χέντς το ανέφεραν. Όντω είναι ζωτική σημασία. Αύριο θα μιλήσετε με τον Δόκτωρ Χέμπροπτ από την Ενίσα και αυτό θα σα πει περισσότερα. Ανανεώσαμε την εντολή τη Ενίσα και τώρα συνεργαζόμαστε μαζί τους προκειμένου να ισχυθεί η συνεργασία στον τομέα του κυβερνοχώρου και της κυβερνοασφάλειας. Εμείς πιστεύουμε ότι με τη συνεργασία στην έρευνα και την καινοτομία μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη και να χρησιμοποιήσουμε έτσι όσο γίνεται καλύτερα και τους εταίρους μας από τις ΗΠΑ. Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα όλοι μαζί, όλα μαζί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να διαθέτουν αυτήν την κυβερνοασφάλεια. Και υπάρχουν διάφορα μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν, αλλά χρειάζεται περισσότερο συντονισμός. Ούτε οι διάφορες, τοπικοί φορείς, ούτε άλλοι έχουν υποστηρίξει μια τέτοια προσέγγιση. Βλέπετε ότι όλο περισσότερο διαβάζουμε στα μέσα ενημέρωσης για τις απειλές αλλά ότι χρειάζεται απάντηση μέσω συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά μεταξύ και επιχειρήσεων και εθνικών αρχών και ευρωπαϊκών αρχών, αυτό είναι κάτι επιπλέον. Ελπίζω το Κοινοβούλιο αυτό θα δει το θέμα με νέα φιλοδοξία. Αυτά όσον αφορά την ασφάλεια του κυβερνοχώρου. Όσον αφορά την νομοθεσία για το ΙΝΤΑ, τώρα δουλεύουμε ακόμα πιο σκληρά όσον αφορά τις εφαρμοστικές διατάξεις. Χρειάζονται ακόμα κάποιες λεπτομέρειες. Το βασικό πρόβλημα του να τα έχουμε όλα ηλεκτρονικά είναι, και νομίζω ότι και οι κοσμήτωρες το ξέρουν αυτό εδώ, εγώ ακόμα πρέπει να υπογράφω πράγματα με το στυλό. Πώς τώρα να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Η Νέλη Κρούς τα έχει καταφέρει, όπως το έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα, αλλά και στο πρόγραμμα του Juncker υπάρχει το ψηφιακό τμήμα στο οποίο αναφέρει τη λέξη οριζόντια. Εμείς μέχρι τώρα λειτουργούσαμε πιο πολύ κάθετα. Υπήρχε ένας αντιπρόεδρος ο οποίος ήταν αρμόδιος. Τώρα όμως, το όραμα για την επόμενη θητεία είναι η ψηφιακή διάσταση να υπάρχει παντού, οριζόντια. Και πράγματι, εγώ δεν βλέπω γιατί να μην είναι προτεραιότητα η ψηφιακή διάσταση παντού. Και τέλος, ερώτηση Κάρεντς, γιατί δεν ε, αγοράζουν μαζικά online οι καταναλωτές. Ότι στις διάφορες δημοσκοπήσεις οι πολίτες φοβούνται. Το ένα, μήπως υπάρξουν απάτες όσον αφορά την πληρωμή τους. Έρχομαι εδώ πάλι στην ασφάλεια του κυβερνοχώρου. Και το δεύτερο είναι ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη ότι αν το προϊόν που θα παραλάβουν δεν τους ικανοποιεί, δεν θα μπορέσουν να το στείλουν πίσω. Πάντως όλο και περισσότεροι αγοράζουν online. Όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν ε, πουλάνε online όλες, ίσως πρέπει και εδώ να φροντίσουμε να τις διευκολύνουμε. Μην ξεχνάτε ότι οι επικεφαλείς πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι τόσο πολύ γνώστες της ψηφιακής τεχνολογίας και πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο κάνουν business. Ίσως θα έπρεπε να μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Ήδη έχουμε στην Ισπανία δύο ε, περιοχές που έχουν επιλεχθεί με ένα σύστημα voucher για να μπορούμε να βοηθούμε επιχειρήσεις. Δηλαδή δίνουμε από 500 μέχρι 5.000 ευρώ, δεν χρειάζεστε και 5 εκατομμύρια. Και έτσι μπορεί κάποια επιχείρηση να ζητήσει τοπικά βοήθεια για να μπορέσει να πουλήσει online. Ελπίζω με τα σχόλια αυτά να απάντησα στα βασικά, στις βασικές σας ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερος γύρος ερωτώ απαντήσεων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και για να ανάψουν λιγάκι τα αίματα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα ήθελα εγώ να δείξω το θέμα του κυβερνοεγκλήματος. Και ε, πρέπει να σας πω ότι αν δεν υπήρχε η δική μας η απόφαση να διαθέσουμε τα 250 εκατομμύρια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα είχε τη δυνατότητα να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Και χαίρομαι που το αναγνώρισε αυτό επιτέλους το καλοκαίρι. Και έχω και ένα διαρθρωτικής φύσεως ερώτημα. Δείξατε ένα βασικό θέμα που έχει σχέση με τις υποδομές και τη σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την αυτονομία των κρατών μελών. Και θέλω να ρωτήσω, αυτά τα περιορισμένα κονδύλια από το Connecting Europe και από το ψηφιακό θεματολόγιο πώς προτιθέμεθα να τα χρησιμοποιήσουμε στη Γερμανία ας πούμε αν θέλουμε να φτάσουμε ε, στο σημερινό επίπεδο της Νότιας Κορέας, τα 50 MB, τότε αυτό σημαίνει 80 δις ευρώ. Και έτσι λοιπόν και τα κράτη-μέλη, αλλά και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση η πραγματικότητα είναι αυτή ότι αυτό μπορεί να γίνει ως επένδυση μόνο από την ιδιωτική οικονομία. Πώς εξελίσσονται λοιπόν οι συζητήσεις και ποια μπορεί να είναι αυτή η μόχλευση που μπορεί να προκύψει σε σχέση με τη χρηματοδότηση. Γιατί όπως ε, σας είπα, ε, τουλάχιστον για το ιδιωτικό τομέα, αυτή η επένδυση μπορεί να γίνει και εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ρικέτ. Ο κύριος Ρικέτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Διευθυντά, θα είμαι σύντομος. Έχω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Και εσείς και πολλοί από εμά υπογράμμισαν το θέμα των επενδύσεων και των υποδομών, πόσο σημαντικό είναι. Έχουμε νέα οικονομικά μέσα, σε συνεργασία βέβαια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για να γίνουν επενδύσεις ακριβώς και, βάση και στη, στα πλαίσια μάλιστα του Connecting Europe Facility, της διευκόλυνσης αυτής. Είμαστε βέβαια σε πειραματικό στάδιο για το 2014 και 2015. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε κατά πόσο υπάρχουν σχέδια ψηφιακών υποδομών που να έχουν μπει στο αυλάκι των ομολόγων έργου και αν ναι, γιατί ποσά. Επίτα μπορείτε να μας εξηγήσετε παρακαλώ γιατί περιορίσαμε, βέβαια το Σεβούλιο κυρίως και εκτός Κομισιόν, την μόχλευση για νέα οικονομικά μέσα, στα πλαίσια πάντα της διευκόλυνσης αυτής για την ε, διασύνδεση στην Ευρώπη. Κυρία Τόγια. Ευχαριστούμε κύριε Διευθύντα για την εισήγησή σας και για το ότι είστε ανοιχτό να εξετάσετε και άλλα θέματα. Η δική μου ερώτηση είναι ε, πολύ πρακτική και συγκεκριμένη αν θέλετε και αφορά στη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ε, τα λίγα κονδύλια σε σχέση με αυτά που είναι απαραίτητα, τα λίγα λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν αρκούν αυτά για να καλύψουμε τις ανάγκες των επενδύσεων. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη και, την, ε, τις, ε, την τοπική αυτοδιοίκηση να χρησιμοποιήσουν σωστά αυτά τα κονδύλια. Αναφερθήκατε στις ε, επενδύσεις, ε, στις ψηφιακές υπηρεσίες. Εγώ τα προσέφτα και ψηφιακές θέσεις απασχόλησης. Να δούμε λοιπόν τι μπορεί να γίνει και θα θυμάστε ότι το Κοινοβούλιο ήταν εκείνο που προσέθεσε αυτή την προτεραιότητα στα πρώτα σχέδια της Επιτροπής. Δεν υπήρχαν τότε τέτοιου είδους θέματα, εμείς τα προσθέσαμε. Άρα δηλαδή καταλαβαίνετε ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια για την περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι αλήθεια ότι από το 4 και το 5 περάσαμε στο 6, θα φτάσουμε και στο 9. Υπάρχει όμως ένα θέμα αποτελεσματικής χρήσης των πόρων. Τα προγράμματα τα οποία εφαρμόζονται ε, από τη Γενική Διεύθυνση την Περιφερειακή και από τις αρμόδιες υπηρεσίες πώς αυτά συνδυάζονται με τη δική σας τη γνώση για την πραγματικότητα, για τις ανάγκες, γιατί ξέρετε αν τελικά τα προγράμματα είναι σωστά, εμείς ε, θα σας πούμε εφαρμόσεστα. Εφαρμόστε Και εσείς λέτε, εμείς κατευθύνουμε λιγάκι την κατάσταση. Και ρωτώ, οι σχέσεις ανάμεσα στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη Γενική Διεύθυνση ε, Ψηφιακής ε, Διασύνδεσης, ποιες ακριβώς είναι οι σχέσεις αυτές. Φοβάμαι ότι δεν είναι τέλεια η συνεργασία, υπολείπεται η συνεργασία και γι' αυτό εμείς ως Κοινοβούλιο τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε στην επόμενη Επιτροπή να υπάρχει σε συνδυασμός αρμοδιοτήτων για να επιτύχουμε το αποτέλεσμα που σήμερα δεν εμφανίζεται. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Χένκελ είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, έκανα, πέρασα όλη μου τη ζωή στον κλάδο αυτό και ε, θέλω να το σκεφτώ λιγάκι, να το διαβάσω αυτό το έγγραφο που μας υποβάλλατε. Και υπάρχει και μια ερώτηση που είναι πώς τα πάμε. Διερωτώ με λοιπόν γιατί εστιάζετε την προσοχή σας τόσο πολύ σε θέματα όπως είναι πόσοι πολίτες κάνουν online αγορές ε, ή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε σχέση με το διαδίκτυο και τις επιγραμμικές διασυνδέσεις. Το θέμα είναι όμως αυτό ενδιαφέρει ή να ε, εστιάζουμε περισσότερο σε άλλα θέματα. Και η δεύτερη ερώτηση, ε, νομίζω πάντα πρέπει κανείς να δίνει το καλό παράδειγμα και αναφέρθηκε εδώ το πώς μπορεί ε, το κοινοβούλιο να ζητάει περισσότερα κονδύλια. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποια πρόταση για το πώς ε, μπορούν οι δικοί μας οι κυβερνώντες να δίνουν το καλό παράδειγμα χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο και την ευρυζωνικότητα. Κατόπιν πάω στους στόχους. Πολύ καλό είναι να έχει κανείς ε, στόχους, αλλά δεν ξέρω αν οι στόχοι μας είναι αρκετά φιλόδοξοι. Μας είπαν ήδη ότι σε κάποιους ε, στόχους ε, δεν τα πάμε καλά, όπως ας πούμε το, τον τρόπο και το πόσο συμπληρώνουν οι πολίτες τα ηλεκτρονικά έντυπα των δημόσιων υπηρεσιών στις Ηνωμένε Πολιτείε, στην Νοτιοανατολική Ασία, στην Κίνα. Εκεί τα πράγματα είναι πιο προχωρημένα. Έχουμε εμείς παρεμφερή σχέδια. Η κυρία Γκροστέτ έχει το λόγο. Καταρχάς κύριε Πρόεδρε θέλω να συγχαρώ τον κύριο Μάντλιν για την καταπληκτική δουλειά που κάνει στο ψηφιακό τομέα. Το ερώτημά μου ή μάλλον πιο πολύ παρατήρηση είναι είναι κάτι αντίστοιχο αυτό που είπε η κυρία Τόγια σε σχέση με την αξιοποίηση των διαρθρωτικών κονδυλίων ώστε τα κράτη-μέλη και η τοπική αυτοδιοίκηση να παρακινηθούν ε, να κάνουν επενδύσεις για την ε, καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος που για μένα είναι προτεραιότητα Θα έλεγα ότι υποχρεωτικά ένα μέρος των ανθρωπικών κονδύλιων θα έπρεπε να αντιμετωπίζει ακριβώς το ψηφιακό χάσμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ασφάλειας, της κυβερνοασφάλειας, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την ιδιωτική ζωή. Υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αρχίζουν να ασχολούνται με το θέμα αυτό και σήμερα αντιλαμβάνονται ότι η ανησυχία αυτή, η μέρημνα για την ασφάλεια της ιδιωτικής ζωής μεταξύ άλλων αφορά πιο πολύ, πιο μεγάλους ανθρώπους ηλικία, αλλά και τη νέα γενιά. Η νέα γενιά βέβαια, αυτό που την ενδιαφέρει είναι να είναι παρόντες στο διαδίκτυο. Αυτό ενδιαφέρει τους νέους. Ό,τι και αν συμβεί. Δεν το θεωρούν πρόβλημα. Την ασφάλεια δηλαδή. Το θέμα είναι να είναι παρόντες, το να μιλάνε ο ένας για τον άλλο, ο ένας με τον άλλο. Δεν είναι λοιπόν για αυτού μεγάλο πρόβλημα η ασφάλεια. Υπάρχουν λοιπόν μικρομεσαίες επιχειρήσει που αρχίζουν να ασχολούνται με την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, σε ό,τι αφορά την ιδιωτική σφαίρα και λένε σήμερα αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μήπως έχουμε αργήσει ήδη πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Κάποιες αποθαρρύνονται λοιπόν ε, ΜΜΕ. Πώς μπορούμε επομένως να στηρίξουμε, να ενθαρρύνουμε την καινοτομία στον τομέα αυτό για να αποφύγουμε προβλήματα. Αλλά υπάρχει και ένα πρόβλημα γενεακό θα το χαρακτήριζα. Εσάς σας απασχολεί αυτό το ζήτημα. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, παρακαλώ. Και ο Κύριε Πρόεδρε, ο κύριο Σουλίνιο, έχει πολλά τεχνικά και τεχνολογικά στοιχεία το ψηφιακό θεματολόγιο. Συμφωνώ όμως με όσους ε, υποστηρίζουν ότι ε, πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει δηλαδή ένα οικονομικό και κοινωνικό πρόγραμμα που θα είναι ανταγωνιστικό. Και είναι ένα εγκάρσιο πρόγραμμα, γιατί αλληλεπιδρά με όλα τα μέλη της κοινωνίας και παρέχει τεράστια ε, ευκαιρία για την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Αυτό είναι πάρα πολύ θεμελιώδες. Υπάρχει το ενδεχόμενο, αν εστιάσουμε πολύ στα τεχνολογικά θέματα, να δημιουργήσουμε μια διπλή εξαίρεση, ένα διπλό αποκλεισμό και θα υποφελούνται μόνο αυτοί που έχουν ε, τις γνώσεις και τη δυνατότητα. Υπάρχει επαρκή στήριξη να έχουμε τη σωστή προσέγγιση γιατί το οργανωτικό μοντέλο που έχουμε και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, στην Κομισιό. Δεν νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις. Το ψηφιακό θέμα το λέω πρέπει να αποτελέσει τη βάση και μετά να μιλήσουμε για μηχανία, ενέργεια, έρευνα τι θέλω να πω ουσιαστικά. Μήπως πρέπει να αναδιοργανώσουμε το μοντέλο λειτουργίας και των ίδιων των θεσμικών οργάνων για να αντιμετωπίσουμε και να αξιοποιήσουμε το δυναμικό αυτού του ψηφιακού θεματολογίου και τις δυνατότητες μας προσφέρει. Συμφωνώ σε ό,τι αφορά την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ή των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι μπορεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει πολλά. Έχω ένα ερώτημα προς τον Ρόμπερτ που είναι και σε καλύτερη θέση από όλου για να απαντήσει, γιατί ήταν και Γενικό Διευθυντής τη ΣΑΝΚΟ, για την ηλεκτρονική υγεία συγκεκριμένα. Βλέπω αυτό το έντυπο, αυτό το τετρασέλιδο και μιλάτε για την επίτευξη των στόχων του ψηφιακού θεματολογίου που θα οδηγήσει σε καινοτόμε υπηρεσίε όπω το e-health, την ηλεκτρονική κτλ. Εγώ θεωρώ ότι είναι κομμάτι ε, του ψηφιακού θεματολογίου. Τι πιστεύετε. Επίσης λέτε να είμαστε φιλόδοξοι και φρέσκοι, να δώσουμε μια νέα πνοή. Τι πρέπει να γίνει για να το πετύχουμε αυτό. Τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. και πάνω στο δικό μας το πεδίο αρμοδιοτήτων. Πώς μπορούμε την ηλεκτρονική υγεία να την προωθήσουμε. Γιατί είναι ένας τομέας που νομίζω δεν έχουμε σημειώσει ακόμη επαρκή πρόοδο. Δεν μιλάω για στόχους, μιλάω για φιλοδοξία. πρέπει να μειώσουμε δραστικά το κόστος στην υγεία, μεν, αλλά ταυτόχρονα να διευκολύνουμε και τη ζωή των πολιτών. Ευχαριστώ. Μπάουλ. Είναι παρόν ή όχι. Δεν είναι πλέον στην αίθουσα. Κυρία um, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον Διευθυντή για την παρουσίασή του, λέει κυρία Νταλή. Υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό που βρήκα στο φυλάδιο που μας δώσατε. Λέτε ότι για να βρει κανείς, ε, μάλλον ότι 6 εκατομμύρια παραπάνω το 2020 θα είναι θέσει απασχόλησης που θα πετούν γνώσεις πληροφορικής. Εσείς τι κάνετε ώστε να υπάρξει η προσφορά για τη ζήτηση αυτή. Τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει τόσο μεγάλη ανεργία, κυρίως στους νέους. Θέλω λοιπόν να ξέρω, εσείς πώς θα βοηθήσετε να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις εκείνες όπου χρειάζεται προσωπικό με γνώσεις πληροφορικής και δεν υπάρχει τώρα. Έρχομαι επίσης στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Το έχουμε εδώ και καιρό. Αλλά αν δει κανεί τόπου τι γίνεται, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν επιχειρήσει που δυσκολεύονται να πουλήσουν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Και υπάρχουν και καταναλωτέ οι οποίοι δυσκολεύονται να αγοράσουν υπηρεσίε ή προϊόντα από άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Πείτε μου λοιπόν, πώ θα διασφαλίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε θα μπορούν να πουλούν τα προϊόντα του και τις υπηρεσίες τους σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και πώς οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες από όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κυρία Σπυράκη έχει τώρα τον λόγο. thank you very much. I am very new here. thank Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Γενική Διευθυντά για την παρουσίασή σας. Ένα σχόλιο έχω να κάνω για το τι χρειαζόμαστε όσον αφορά την ενιαία ψηφιακή αγορά. Θέλω να σας ρωτήσω, πρέπει να αρχίσουμε από το α μικρό, γιατί όταν ανταγωνιζόμαστε με τις ΗΠΑ Πολιτείες η Ευρώπη πρέπει να έχει πλεονεκτήματα. Τον έχουμε 20 διαφορετικές ε, αγορές βάσει των εθνικών συνόρων δεν βοηθάει. Και <clears throat> η εμπορία στην Αμερική είναι πολύ πιο εύκολη γιατί έχουν 300 εκατομμύρια καταναλωτές εκεί και είναι ενιαία αγορά. Αν λοιπόν ήταν μια ενιαία αγορά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαμε να αποφεληθούμε από 500 εκατομμύρια ε, καταναλωτές το διπλό σχεδόν από αυτό που έχουν, που έχει οι ΗΠΑ σήμερα. Πρέπει να βιαστούμε λοιπόν, πρέπει να ξεπεράσουμε τι αντιστάσει των χωρών μελών και να φροντίσουμε να μην χάσουμε τις ε, θέσεις αυτές που θα μπορούσαμε αλλιώ να έχουμε κερδίσει στο εμπόριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Πέρες μόλις βγήκε. Φαντάζομαι θα επιστρέψει. Ο κύριος Ετσενίκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαντελέν που ήσασταν εδώ σήμερα. Δεν έχω καμιά αμφιβολία για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να λύσει τα προβλήματα ηλεκτρονικού εμπορίου κτλ. Εγώ στι ΗΠΑ αγόρασα ε, στο Amazon από μια ισπανική εταιρεία. Άρα τα σύνορα δεν είναι και τόσο πολύ εμπόδιο για τις ψηφιακές αγορές αλλά θέλω να αναφερθώ σε ένα σημείο που νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο από αυτό. Και αυτό είναι οι υπολογιστέ, το κυρίως κομμάτι των υπολογιστών που κάνει την επεξεργασία. Νομίζω ότι σε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται πολύ πίσω σε σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Φαίνεται επίσης ότι χρειάζεται μια βιομηχανία πολύ περισσότερο επικεντρωμένη στην έρευνα για να μπορέσουμε να καλύψουμε τη διαφορά. Θέλω λοιπόν να ξέρω τη δικιά σας τη γνώμη. Υπάρχει κανένα σχέδιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου η Ευρώπη να ευθυγραμμιστεί με τις ΗΠΑ ακόμα και με την Κίνα που από φαίνεται πάει όλο και πιο γρήγορα στο θέμα αυτό τη επεξεργασία δεδομένων. Είναι ζωτική σημασία, πιστεύω, το θέμα αυτό του φτιαξίματο των υπολογιστών, της κατασκευής. Ευχαριστούμε κυρία Κάπελ. Αξιότιμε Πρόεδρε, κύριε Γενική Γραμματέα, σήμερα στο πλαίσιο της ε, γενικότερη συζήτηση για τον προπλογισμό ακούσαμε ότι υπάρχει χρηματοδοτικό κενό του 10% ε, στην έρευνα και την ανάπτυξη και αυτό το κενό, το έλλειμμα ε, προφανώς επηρεάζει και το ψηφιακό θεματολόγιο. Εσείς ο ίδιος κύριε Γενική Διευθυντά είπατε σήμερα ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ιδιωτικές επενδύσεις για την επέκταση των υποδομών. Και ερωτώ, η Γενική Διεύθυνση, η Επιτροπή να λάβει μέτρα έτσι ώστε να προσελκύσει περισσότερους επενδυτές για αυτές τις υποδομές και αν ναι πια ακριβώς ε, μήπως πρόκειται να υπάρξει και συνεργασία με άλλες γενικές διευθύνσεις γιατί αν κατάλαβα καλά από αυτά που μας είπατε αυτό που σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι να προσελκύσετε ιδιώτες επενδυτές. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μάρτιν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο. Θέλω απλώ να επιστήσω την προσοχή του προσκεκλημένου μα στη στάση τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε σχέση με τα διάφορα προγράμματα που, στα οποία επενδύει. Κινδυνεύει να χάσει το τριπλό Α. Μερικές φορέ έχει και μια στάση όπως οι ιδιωτικές επενδυτικές εταιρείες. Κάτι το οποίο βέβαια αποτελεί τροχοπέδι για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και περιορίζει τις επενδύσεις. Μια που δεν ηγείται των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνειδητοποιεί τον ρόλο αυτό της ε, ΕΠΕ που περιορίζει τελικά τις επενδύσεις και κάνει κάτι προκειμένου η ΕΤΕ να μπορέσει να παίξει πλήρω το ρόλο της σήμερα μάλιστα που είμαστε σε ευρωπαϊκή οικονομική κρίση χωρίς άλλο προηγούμενο. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω άλλο στον κατάλογό μου. Η κυρία Μπέρες δεν είναι εδώ, ε. Δεν είναι στην αίθουσα. Ωραία. Να ακούσουμε την απάντησή σας τότε. Οι ερωτήσεις ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσε. πιστεύω και λεπτομερείς, οπότε εμείς περιμένουμε τώρα να μας απαντήσετε, να σταθείτε στο ύψος. Αυτό περίμενα ότι θα μου λέγατε. Καταρχάς να συνδέσω αυτό που είπε ο κύριος Μαρτά με τις ερωτήσεις των κύριων Χέγκελ και Ρουκέ στην αρχή. Διότι όλα μιλούν για τα ομόλογα έργων, πώ ε, η ΓΔ Connect, το τηλεπικοινωνικό σκέλο, ε, η IB, ε, πώς όλοι αυτοί συνεργάζονται. Να ξεκινήσω με το ερώτημα του κύριου Ρούκη. Αν ε, κάτι έχει μπει στο αυλάκι. Ναι, έχει μπει. Και τι, έχει, ε, τι απομένει να γίνει δεν μπορώ, αλλά μπορώ να σας στείλω ένα email με τις λεπτομέρειες αργότερα. Δεν έχω ενημερωθεί μετά το καλοκαίρι. Αλλά, και τώρα στρέφουμε στο ερώτημα του κύριου Μαρτά, η εντύπωσή μου είναι ότι τα μέλη της ομάδας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων έχουν στόχους, ε, όπως ε, κάθε καλός ε, εργαζόμενος. Κάποιες φορές όμως υπάρχουν διαφωνίες, διαφορετικές προσεγγίσεις. Οπότε ή κάποιος πρέπει να αναλάβει ρίσκο και μια σειρά μικρών προγραμμάτων μπορεί να μην είναι η βασική δραστηριότητα. Και έπειτα έχουμε και το επίπεδο των συμβουλίων, το Διοικητικό Συμβουλίο έχει κάνει πολλά η Νέλη Δεν θέλω ε, να μιλήσω υπέρ κατά το τραπεζών. Νομίζω ότι προχωρούμε προς πιο καινοτόμες προσεγγίσεις, αληθεύει όμως ότι το τίμημα θα είναι μεγάλο. Αν μπορούμε να έχουμε επιτυχημένα πιλωτικά προγράμματα μέσα στα επόμενα ένα-δύο χρόνια, νομίζω ότι στην διάμεση αξιολόγηση, αναθεώρηση θα ξαναδούμε το θέμα της χρήσης των δημοσίων κονδυλίων ε, με ε, αποτελεσματικό τρόπο για να έχουμε μόχλευση ε, και ιδιωτικών επενδύσεων. Και η θετική συμβολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων μέσω των πιλωτικών προγράμματων θα είναι πολύ πιο σημαντική από ό,τι μέχρι τώρα. Αυτή λοιπόν είναι η απάντησή μου. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν και δύο άλλα πράγματα, διαρθωτικά ταμεία και ρυθμιστικό πλαίσιο, έπιασαν και σχολίασαν και άλλοι συνάδελφοι τα σχετικά. Η κυρία Τόγια και τα διεθνωτικά προγράμματα είπε τώρα που ε, Έχουμε εσωτερική συνεργασία. Ναι, πράγματι υπάρχει συνεργασία. Δεν είναι τέλεια βέβαια και προσπαθούμε να την βελτιώσουμε. Στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ οι συνάδελφοί μου, αλλά και σε μια άλλη ομάδα, JIC, για την ευφύ εξειδίκευση και οι συνάδελφοι από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Απασχόληση που εξετάζουν τις δεξιότητες, η ομάδα για τις ΜΜΕ, στη ΓΑΜΑ επιχειρήσεις, όλοι αυτοί ε, προσπαθούν από την ίδια πίτα αν θέλετε να πάρουν κάτι αλλά να βελτιώσουν ουσιαστικά τα πράγματα και όπως ε, είπε και ο κ. Ζουνίου ε, πρέπει να συνεργαστούμε καλύτερα, να οργανωθούμε καλύτερα και πράγματι υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται ακριβώς με αυτό το θέμα τώρα που μιλάμε. Ελπίζω πάντως ο τρόπος για να επιτύχουμε την αλλαγή να αλλάξουμε τι απαιτήσει των δικαιούχων. Να όλοι οι δήμαρχοι, οι περιφερειακοί σύμβουλοι, όλα τα κράτη-μέλη τακτικά σε διάφορους υπουργούς ή σε ε, διάφορους υπεύθυνους για την οδοπία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλαζαν την προσέγγισή τους, θα άλλαζε και η ανταπόκριση σε ό,τι αφορά το στόχο της συγκέντρωσης στον τομέα των επικοινωνιών. Δεν θα έχουμε διπλή συγκέντρωση ICT στον προγραμματισμό, αλλά με την Επιτροπή των Περιφερειών, την Οικονομική Επιτροπή, με εσά, ε, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ήδη από αυτό το μήνα μπορούμε να ξεκινήσουμε κάποια σχέδια, πλαίσιο και να προσδιορίσουμε καλύτερα του στόχου μα. Και τι είναι αυτοί οι στόχοι. Θέλουμε ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων από το δημοτικό μέχρι το τέλο ε, τη ε, υποχρεωτική εκπαίδευση και σε όλη τη διάρκεια τη επαγγελματική σταδιοδρομία. Θέλουμε να βελτιώσουμε τι δεξιότητε και των επιχειρηματιών. Επανέρχομαι στον κύριο Κάριν να παράσχουμε τοπική βοήθεια, δηλαδή βοήθεια σε τοπικό επίπεδο. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τη βοήθεια που μπορούν να παράσχουν ε, όσοι, έχουν, ε, όσοι τα καταφέρουν καλύτερα στον τομέα αυτό και να βοηθήσουν αυτούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και ποιο θα μπορούσε να είναι το τοπικό ψηφιακό θεματολόγιο. Νομίζω ότι με την, υψηλή, με την ε, ευφυή εξειδίκευση αρχίζουμε λίγο να βλέπουμε κάποια αποτελέσματα. Είναι πολύπλοκος ο τομέας, πράγματι θα χρειαστεί χρόνος. Με τη βοήθειά σας ελπίζω να καταφέρουμε πάντως. Για τους κανονισμούς, για τις ρυθμίσεις, ε, το TSM σίγουρα δεν είναι το τέλος Ελπίζω ότι είναι επιτάπητο να το ολοκληρώσουμε πάντω, γιατί αυτό θα είναι σημαντικό, ιδίω ό,τι αφορά την περιαγωγή, για παράδειγμα, που είναι ένα πολύ ορατό πρώτο επίτευγμα, ελπίζω, το Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά δεν αρκεί, πρέπει να γίνουν και άλλα. Και θα τα συζητήσουμε και φαντάζομαι με τον κύριο Γιούγκερ και τη νέα επιτροπή μετά την αλλαγή σκητάλη. Χένκελ τώρα. Για τους δείκτες επιδόσεων, ε, πολύ καλό το ερώτημά σας. Για το 2010 βάλαμε κάποιους δείκτες που θεωρούσαμε ότι ήταν σημαντικοί ή ενίοτε βάζουμε στοιχεία που έχουμε. Γι' αυτό και επιλέγουμε συγκεκριμένους δείκτες. Σίγουρα καλό θα ήταν να βελτιωθούμε. Και όταν αλλάξει η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα επανεπικυρωθεί το ψηφιακό θεματολόγιο και εκεί θα δούμε ποια είναι τα πέντε πράγματα που μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Και να δώσω και απάντηση στο ερώτημά σας για τον αντίκτυπο. Ένα δεύτερο ερώτημα που θέσατε ήταν σε ποιους τομείς μέχρι τώρα έχουμε ξεκινήσει να δίνουμε, αν θέλετε, το καλό παράδειγμα. Θέλετε ίσως να ευλογήσουμε τα γένια μας. Δεν με... Ποτέ δεν μου αρέσει να το κάνω αυτό, αλλά τέλος πάντων υπάρχει ένα παράδειγμα με αυτούς τους δείκτες αντικτύπου. Εάν δείτε ε, τι συνδέσεις, τι links έχουμε στην, ε, στο φυλάδιο αυτό, θα δείτε σε μία από αυτές τις συνδέσεις αναλυτικά ε, τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων μας, γιατί νομίζουμε ότι πρέπει να αναλαμβάνουμε ευρωπαϊκά αυτές τις δράσεις, τι πόρους έχουμε διαθέσει σε κάθε δραστηριότητα και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Αν θέλετε λοιπόν να εμβαθύνετε και ίσως θα μπορούσατε μετά να μας δώσετε και κάποια μηνύματα, να μας πείτε ότι αυτό δεν είναι σημαντικό, σε αυτό πρέπει να δοθεί περισσότερη πόρη κτλ. Μπορούμε να επικαιροποιήσουμε, το επικαιροποιήσαμε ε, τον Ιούλιο ε, το φυλάδιο, αλλά σίγουρα μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμη τα πράγματα. Και κάτι άλλο. Θα έχουν σε ταμπλέτα την, ε, το briefing τους την επόμενη φορά, μην τους το πείτε ακόμα. Και τρίτον, με τους ε, συναδέλφους από τη ΓΑΜΑ ΜΑΡΚΤ, θέλουμε να είναι ταχύτερο το e-procurement στην Κομισιόν. Θα θέλαμε να γίνονται οι διαγωνισμοί ηλεκτρονικά σε μεγαλύτερο βαθμό. Για την κυρία Γκροστέτ, χρησιμοποίησατε τη λέξη εμποζέ, επιβάλλω. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι που μπορεί να το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα, αλλά σίγουρα ε, μέχρι στιγμής σταματάμε στη μέση. Λέμε να έχουμε ένα στόχο συγκέντρωσης, αλλά περιμένουμε να συμφωνήσουν όλοι για να το επιτύχουν. Σίγουρα βάζουμε ένα στόχο, αλλά δεν τον επιβάλλουμε τόσο πολύ αν θέλετε δεν είμαστε τόσο αποφασιστικοί. Αν κάποια κράτη-μέλη δεν το παίρνουν πολύ καλά, φανταστείτε τι θα νιώθουν κάποιοι πάλι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σίγουρα μπορούμε να είμαστε πιο καθοδηγητικοί. Και έρχομαι στην οδηγία για το NIS. Μπορούμε να ζητήσουμε από τις εταιρείε όταν έχουν μια κυβερνοεπίθεση να συνεργάζονται με τις κυβερνήσεις και οι κρατικοί φορείς μπορούν ε, να υποχρεωθούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες με άλλες χώρες που είναι υπό απειλή. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ε, κατοχυρωθεί στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Άρα είναι θέμα του πόσο σκληρά προσπαθούμε και είναι ένα πολιτικό ζήτημα μείζον. Και έχει να κάνει και με το επενδυτικό χάσμα. Το ψηφιακό θεματολόγιο είναι μόνο λόγια ή μπορούμε να έχουμε και αποτελέσματα. Επίσης, κύριε Γκροστέτ, με ρώτησε αν έχω κάποια ε, άποψη σε ό,τι αφορά ε, τη θέση που έχουν οι νεότερες και μεγαλύτερες γενιές ό,τι αφορά την κυβερνοασφάλεια. Μπορώ μόνο να φανταστώ τι μπορεί, να διαισθανθώ τι μπορεί να νιώθουν νεότεροι, αλλά υπάρχει αλλαγή νοτροπίας σε κάθε γενιά, γιατί έχει να αντιμετωπίσει τα νέα αυτά εργαλεία, ανταποκρίνεται και κάθε γενιά ανταποκρίνεται διαφορετικά. Μετά από 5-6 χρόνια αλλάζει η στάση μας και η αντιμετώπιση μας. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορεί να ήταν cool και δεν είναι πλέον πραγματικά για τη 12χρονη ανιψιά μου. Αλλά είναι και θέμα να κατανοήσει κανείς όρημα τι μπορεί ε, κάποιος να κάνει αν δεν είναι διακριτικός. Παραδείγματο χάρη, ε, επειδή ανέβασα στο διαδίκτυο κάποιε φωτογραφίε από ένα περσινό πάρτι, χάνω μια δουλειά. Ε, δεν την παίρνω τέλο πάντων. Υπάρχουν ατυχή συμβάντα, αλλά δεν προέρχονται αυτά μόνο από τους νέους. Υπάρχουν κάποιοι μεγαλύτεροι ηλικία που κάνουν αρκετές ανοησίες και στο διαδίκτυο και δεν μιλώ μόνο για ε, κάποιες οικονομικές αλλά και για selfies που μπορεί να πάρουν. Δεν νομίζω όμως ότι οι νέοι δεν θέλουν ε, την ιδιωτικότητα. Το αντίθετο θα έλεγα. Αλλά μιλάμε για μια βιώσιμη αϊφόρο κατανάλωση. δεν έχει υπάρξει ακόμη αρκετή ζήτηση από αυτούς οι οποίοι ε, είναι συνέχεια στο διαδίκτυο για μεγαλύτερη ασφάλεια. Μας ενδιαφέρει να αγοράσουμε ένα φθηνό προϊόν. Για το ερώτημα του κ. Ταλίτσκη, συμφωνώ για την υγεία, η ηλεκτρονική υγεία ότι είναι μέσα στο ψηφιακό θεματολογείο, είναι Έλλη και ο αρμόδιος για την υγεία επίτροπος είναι υπερήφανη για τη συνεργασία που είχαμε, για την ενεργογύρανση. Πώς μπορούμε την υγεία, την ψηφιακή υγεία να την ε, προωθήσουμε καλύτερα. Πρώτον, με, τις, με την αλληλεπίδραση που έχουμε με τις οικονομικές υπηρεσίες, θα πρέπει κάθε γιατρός να πιστεί τα δεδομένα του ασθενούς να τα αντιμετωπίζει ακριβώς ως τέτοια και όχι δεδομένα που έχει αυτός στη διάθεσή του. Υπάρχει ε, ένα σύλλογο ε, δέκα χρόνια έκλεισε και ήμουνα στην εκδήλωση που έκαναν γι' αυτό. Είναι σημαντικό να δείχνουν ε, στον ασθενή όταν του λένε τα αποτελέσματα κάποιων εξετάσεων, εικόνες από τον υπολογιστή τους, οι γιατροί. Επίσης, ανωνυμοποιημένα δεδομένα για υγεία. Αν βάλω το γονιδίωμά μου δίπλα στο γονιδίωμα ε, του κυρίου βουλευτού, υπάρχουν κάποια ηθικά θέματα. Ε, πώς μπορούμε να επιτρέψουμε μια ανάμειξη δεδομένων. Δεν θέλω να έχει Ιατρική Επιτροπή ε, πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία ή αρμόδια υπηρεσία της Κομισιόν. Αν όμως τα στοιχεία μου ε, τα αναμίξω με τα στοιχεία όλων εδώ στην αίθουσα, μπορώ να σώσω ζωές, τι κάνω σε αυτή την περίπτωση. Δεν τα έχουμε ξεκαθαρίσει όλα αυτά. Επειδή πάντα υπάρχει ένας ασθενής και ένας γιατρός, η συγκατάθεση είναι εύκολη να επιτευχθεί, αλλά τώρα τα έχουμε όλα ηλεκτρονικά και δεν γίνεται αυτό αυτή η επικοινωνία. Οι ερευνητές το της υγείας μας λένε ότι δεν είναι σίγουροι ότι έχουν ε, προχωρήσει αρκετά τα πράγματα. Θα δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα της ε, ηλεκτρονικής υγείας. Και για τα τρία λεπτά που μου απομένουν έχω να απαντήσω δύο ερωτήματα. Νταλή και Σπυράκη, οι δύο κυρίες έθεσαν ενδιαφέροντα ερωτήματα παρόμοια. Χρησιμοποίησαν ε, παρόμοια διατύπωση. Έχω μια αγορά 500 εκατομμυρίων. Δεν υπάρχει μια δυσπόζουσα γλώσσα, ούτε δύο θα έλεγα. Ε, Όπω ισχύει με τη ΣΥΠΑ για παράδειγμα. Έχουμε ένα πρόβλημα γλωσσικό. Θα πρέπει επομένω να συνεχίσουμε να επενδύουμε στις, στην καινοτομία σε ό,τι αφορά ε, τις ε, μεταφράσεις από μηχάνημα. Πρακτικός είναι ο λόγος βέβαια. Και πρέπει να επενδύσουμε. Και σε αυτό, αλλά είπα και άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν, να ένιωσε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ο καταναλωτής. Μίλησε σχετικά και ο Ένα είδος Advisor. Μπορούν να δημιουργηθούν κάποιε μηχανέ που θα βοηθούν του καταναλωτέ, να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο ποιο πάροχο υπηρεσιών είναι καλός πέραν των πολύ γνωστών και μεγάλων. Τέλο πάντων, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα χωρίς πολύ μεγάλο κόστος. Επανε... Επανεκβιομηχάνηση, Πολύ σημαντικό θέμα. Για τα τσίπς, για τα ενσωματωμένα συστήματα έχουμε μερίδες στην αγορά. Αλλά ιδιωτικές συμπράξεις που προανέφερα για όλα αυτά τα στοιχεία, φωτονική κτλ. Στόχο έχουν να δημιουργήσουν εκ νέου μια βιομηχανική βάση. Με τη χρηματοδότηση ε, από το 2020 στις επόμενες χρονιές θα βελτιωθούμε στους τομείς αυτούς. Και α, για το σχόλιο της κυρίας Κάπελ για την ευρωζωνικότητα νομίζω το, κατέλη, ε, το, το συζήτησα. θα έχουμε ένα πρόβλημα 150 εκατομμυρίων φέτος. Θα πρέπει να τα βγάλω το 2015 να πληρώσω και τόκους. Και μειώνονται και οι πιστώσεις πληρωμών. Είμαστε στην κατάσταση που ήταν και περισσότερες ευρωπαϊκές μοναρχίε του 17ου αιώνα. Πτωχεύσει, ε, τέλο πάντων μήπως δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω αυτή την ε, παρομοίωση. 35 χρόνια που είμαι υπάλληλος δεν το έχω ξαναβιώσει, και είναι πολύ δύσκολο ε, και θα γίνει και χειρότερα το 2015. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Το ψηφιακό θεματολόγιο είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει κατά προτεραιότητα τους επόμενους μήνες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό που το συζητήσαμε σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και σας ευχαριστώ και σας όλους για τις ερωτήσεις σας. Ο κύριος Μάρβιν ακόμα εδώ μαζί μας και ο κύριος Μεντελίν αξίζουν πιστεύω ένα γερό χειροκρότημα. Ωραία, περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι και το τελευταίο θέμα μας για σήμερα. Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή 2014, COP20, στην Λίμα του Περού. Εξετάζουμε, ανταλλάσσουμε απόψεις για ένα σχέδιο γνωμοδότησης. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, αγαπητοί φίλοι, φεύγετε. Αυτό βέβαια μας απασχολεί, αλλά είναι δικαίωμά σας, το ξέρω. Σας παρακαλούμε όμως όσοι φεύγετε από την αίθουσα να το κάνετε ησύχως γιατί εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Λοιπόν, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας αλλά και της Επιτροπής Περιβάλλοντος θα πάνε στην διάσκεψη αυτή των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στη Λίμα του Περού. Ετοιμάζοντας λοιπόν τις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν εκεί, ετοιμάζουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ψήφισμα. Μου ζητήθηκε λοιπόν από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ήτρε να ετοιμάσω εγώ κάτι που να αποτελεί τη δικιά μας συνεισφορά στο σχέδιο ε, ψηφίσματος που ετοιμάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Γιατί το τελικό ψήφισμα είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Περιβάλλοντος, της ΕΝΒΗ. Αλλά και εμείς θέλουμε να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις. Γενικά μιλώντας λοιπόν, είναι σαφές ότι η επιτυχία της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, είναι ένα συλλογικό θέμα. Πρέπει να υπάρξουν συλλογικές δράσεις για να το πετύχουμε. Η Ευρώπη ξέρουμε ότι θέλει να έχει ηγετική θέση στον κόσμο επ' αυτού. Όμως όλες οι χώρες πρέπει να συνεισφέρουν για να περιοριστούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Για να περιοριστεί η κλιματική αυτή αλλαγή που αποτελεί μία απειλή. Δεν είναι όπως η όξινη βροχή που ήταν καθαρά τοπικό φαινόμενο. Αυτό εδώ, η αλλαγή κλιματική, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Συνεπώς έχουμε την ε, ευκαιρία με τη διάσκεψη αυτή να προχωρήσουμε για περισσότερη ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη. Αλλά όπως είπαμε είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει ολόκληρο τον πλανήτη και όχι να προέρχονται οι πρωτοβουλίες μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση το σχέδιο του ψηφίσματος αυτός χωρίζεται σε τρία τμήματα. Το πρώτο είναι η βιομηχανία και η ανταγωνιστικότητα, το δεύτερο είναι η έρευνα και η καινοτομία και το τρίτο είναι η ενεργειακή πολιτική. Για το πρώτο τη βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητα. Τεχνολογικά μιλώντας, η Ευρώπη είναι πολύ σημαντική όσον αφορά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Οι αγορές όμως κατά τη γνώμη μας, και αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί ως παρατήρηση στο ψήφισμα, οι αγορές πρέπει να επιτρέπουν την ε, εισαγωγή ε, φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών και να μην ε, υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Έρχομαι τώρα στην έρευνα και την καινοτομία. Εδώ θέλουμε φυσικά να έχουμε ηγετική θέση. Το θέμα είναι όμως ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ιαπωνία, αλλά είναι πολύ σημαντικό και για μας, ε, οι χώρες αυτές είναι αρκετά προηγμένες, γι' αυτό χρειάζεται συνεργασία με όλους τους διεθνείς εταίρους μας. Και το τρίτο θέμα, ενεργειακή πολιτική τώρα. Η ενεργειακή πολιτική απαιτεί επίσης διεθνή δράση για να αποφύγουμε την εξωτερήκευση του κόστους και για να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος μέσω των κατάλληλων εμπορικών προγραμμάτων όσον αφορά τις εκπομπές αυτές. Και είναι κρίμα που δεν, υπάρχουν, ε, δεν υπάρχει μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης διεθνώς. Αυτά λοιπόν είναι τα πιο σημαντικά σημεία στο δικό μου το κείμενο. το οποίο, ξαναλέω, θα είναι η συνεισφορά της Επιτροπής μας στο σχέδιο ψηφίσματος που ετοιμάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Υπάρχουν εδώ σκιώδεις οι συγητές που θέλουν ίσως το λόγο από πλευρά των σοσιαλιστών, η κυρία Φαν Μπρέμπτ. Παρακαλώ, κυρία Φαν Μπρέμπτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω πρώτα απ' όλα να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις πριν αναφερθώ στις δικές σας τροπολογίες, λέει η κυρία Το COP20 στη Λίμα το Δεκέμβριο είναι μια πολύ σημαντική διάσκεψη. Πρέπει να δούμε, και είναι αυτό σημαντικό αλλά και δύσκολο, πρέπει να δούμε φιλόδοξους στόχους από όλους τους παίκτες, όχι μόνο από την Ευρώπη, θα επανέλθω σε αυτό αργότερα, και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Κίνα και από τη Ρωσία. Είναι απαραίτητο αυτό αν θέλουμε να πετύχουμε την επόμενη χρονιά στο Παρίσι. Γι' αυτό λοιπόν και ανησυχώ κάπως. Το Σεπτέμβριο τώρα οργανώνει ε, μια διάσκεψη για το κλίμα, ο Μπακιμούν, όπου είναι προσκεκλημένοι όλοι οι ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων. Ελάχιστοι όμως πρωθυπουργοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρευρεθούν. Αυτό κάτι δείχνει για τη σημασία που δίνουν οι πρωθυπουργοί μας σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Η ευθύνη της Ευρώπης είναι ζωτική σημασίας και έχετε και εσείς μια σχετική τροπολογία. Γι' αυτό λέω, είναι πολύ σημαντικό αλλά και ανησυχητικό που ακόμα σήμερα η Ευρώπη δεν έχει ένα δικό της σχέδιο, συζητάει, αλλά δεν έχει τους δικούς της στόχους, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε στις αρχές χρονιάς, πότε ήταν το Φεβρουάριο, ένα πολύ σημαντικό ψήφισμα στο οποίο έλεγε με σαφήνεια ότι θέλει 40% μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, 40% ενεργειακή αποδοτικότητα και 30% εναλλακτικών πηγών ενέργειας και αυτά μέχρι το 2030 η ομάδα μου θα ήθελε να είμαστε περισσότερο φιλόδοξοι, αλλά κάτι είναι και αυτό. Πρέπει λοιπόν αυτοί οι στόχοι να συμπεριληφθούν στο γενικό ψήφισμα. Ξέρω ότι από τη δικιά μας την Επιτροπή θα περιοριστούμε στις δικές μας αρμοδιότητες. Αλλά είναι σημαντικό να φανεί ότι όλες οι ομάδες συμφωνούμε. Έρχομαι τώρα στις δικές σας τροπολογίες. Γενικά μιλώντας, τις στηρίζουμε. Είναι καλές και συνάδουν με τις συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί ως τώρα στην Επιτροπή Ήτρε στην προηγούμενη θητεία. Υπάρχουν τροπολογίε σα 13 και 14, οι οποίε περιλαμβάνουν ένα ιδιαίτερα ισχυρό μήνυμα και συμφωνώ πολύ μαζί του. Αλλά υπάρχει. θα ήθελα να πω για τι τις τροπολογίες 1, 5 και 6 ότι χρειάζονται κάποια διευκρίνηση κάποια διαφορετική ίσω διατύπωση, γι' αυτό και θα υποβάλω κάποιε δικέ μου σχετικά. Κατά τα άλλα και γενικά μιλώντας σα λέω ότι συμφωνώ, είναι πολύ σωστή η προσέγγισή σας. σε ευχαριστούμε πολύ. Επόμενο και συζητητή είναι ο κύριο Φέντερλεϊ από την Άλντε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, γενικά πολύ καλέ οι τροπολογίε σα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε περισσότερο βέβαια ότι Θέλουμε να εξακολουθούμε να έχουμε η οικονομική ανάπτυξη που να αποδεσμευτούν από τον περιορισμό των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θα μπορούσαν να ήταν πιο ισχυρά. Θα επανέλθουμε αργότερα. Πάντως, καλό είναι που αναφερόμαστε στις ΗΠΑ και στην Κίνα η ομάδα μας νομίζω ότι θα πει ότι η αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να είναι να δει ότι και στι Ηνωμένε Πολιτείε και την Κίνα μειώνονται οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Αυτά είναι τα πρώτα μου σχόλια, τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ρότζερ Χέλμερ, που και αυτός είναι εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ μιλώ εκ μέρου της Ομάδας Ελευθερίας και Δημοκρατίας, αλλά πρέπει να σας πω ότι και στη δική μας την ομάδα, ακόμα και σε εμά υπάρχουν διαφωνίες. Νομίζω συμφωνούμε βέβαια όλοι μας ότι αυτό που μας απασχολεί είναι η θέση απασχόληση, οι επενδύσεις και η ανταγωνιστικότητα. Βέβαια για μεγάλο χρονικό διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θέλησε να δώσει το καλό παράδειγμα και υποθέτοντας ότι οι επόμενοι θα ακολουθήσουν. Το πρόβλημα όμως είναι ότι πολύ λίγες χώρες ακολουθούν αυτό το παράδειγμα. Και η Αυστραλία που ξεκίνησε τώρα αλλάζει θέση. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι προκαλέσαμε τεράστια ζημιά στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο κύριος Ταγιάννη, ο απερχόμενος, πρόσφατα είπε ότι έχουμε προκαλέσει στην Ευρώπη βιομηχανική σφαγή με τις τιμές που έχουμε επιβάλει και δύσκολο να διαφωνήσει κανείς μαζί του. Ε, στην Κίνα κατασκευάζονται ε, πυρηνική μάλλον ε, σταθμή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως και στη Γερμανία περίπου 1200 ε, τέτοιου είδου σταθμοί και μια τελευταία μελέτη του Πανεπιστημίου του Πρινστον αναφέρει ότι οι υποχρεώσεις απέναντι σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας από ορυκτά κάψιμα θα αυξηθούν κατά το ε, εγγύς μέλλον. Άρα δηλαδή είναι σαφές οι προσπάθειές μας τελικά δεν, δεν στέφονται από επιτυχία. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, εργασία και επενδύσεις, αλλά αυτά τα διώχνουμε από την Ευρώπη και πολύ συχνά τα οδηγούμε σε άλλα κράτη με χαμηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα. Το αποτέλεσμα είναι ότι εδώ στην Ευρώπη χάνουμε και θέσεις απασχόλησης και ε, επενδύσεις και αυξάνονται μάλιστα και εκπομπές. Δηλαδή χάνουμε από παντού, χαμένοι από χέρι και αυτό δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να το δεχόμαστε. Και επανέρχομαι στην δική σας την έκθεση, στο σχέδιό σας πρόεδρε. Εσείς ε, με βάση αυτά που λέτε, όλα αυτά είναι πολύ ευκταίοι στόχοι, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ενεργειακή επάρκεια, αλλά η εμπειρία έχει δείξει ότι όλα αυτά δεν γίνονται. Η εμπειρία ε, από τις κλιματικές διασκέψεις είναι ότι αποτυγχάνουν αυτές γιατί εμείς στην Ευρώπη μπορεί να θέλουμε να προχωρήσουμε αλλά άλλες χώρες ε, παραμένουν μόνο στις μεγαλοστομίες. Γι' αυτό λοιπόν τουλάχιστον στις συστάσεις μας να συμπεριλάβουμε μία ρήτρα που να λέει ότι ε, ως Ευρώπη δεν θα κάνουμε και εμείς μόνοι μας ε, βήματα που δεν θα ακολουθήσουν άλλες χώρες γιατί αυτό βλάπτει την οικονομία μας. Πρόεδρος, δεν έχουμε άλλον σκιώδη εισηγητή παρόντα. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος να λάβει το λόγο. Από ό,τι βλέπω όχι. Και έτσι λοιπόν θα ήθελα να παρακαλέσω τον εκπρόσωπο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση Κλίματος να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπούζεκ που μου δίνετε τη δυνατότητα να πω λίγα λόγια. Νομίζω στην εισαγωγή σας πολύ σωστά είπατε ότι η συνδιάσκεψη COP20 στη Λίμα θα αποτελέσει ορόσημο ε, στο Παρίσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να επιτύχει μια νέα συμφωνία ανάμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, τα σημαντικά τουλάχιστον. Αν δούμε λοιπόν ε, τις πολιτικές εξελίξεις για την ε, κλιματική πολιτική σε διεθνές επίπεδο, βλέπουμε να υπάρχουν ελπίδες, διότι η κυβέρνηση Ομπάμα στις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει σοβαρά υπόψη της την κλιματική αλλαγή και προσπαθεί να εισάγει κλιματική νομοθεσία στις ΗΠΑ, κάτι που δεν υπάρχει κατά το παρελθόν. Παρεμφερήσει κινήσεις και στην Κίνα. Αυτή τη στιγμή η Κίνα με το σύστημα ανταλλαγής ε, ποσοστώσεων εκπομπών θέλει να ε, προχωρήσει και μετά το 2020. Άρα δηλαδή βλέπετε υπάρχουν χώρες που ακολουθούν το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν είχαμε την τελευταία μας συνάντηση τον Ιούνιο και οι υπουργοί μας σε διεθνές επίπεδο έπεισαν τους υπόλοιπους ότι μπορεί κανείς και να ε, επιτυγχάνει την ανάπτυξη της οικονομίας του και να περιορίζει το ε, αποτύπωμα άνθρακα. Κατά το παρελθόν, ένα από τα επιχείρηματα που αναφέρονταν ήταν ότι είτε θα αντιμετωπίσει κανείς τη φτώχεια είτε την κλιματική αλλαγή. Όμως σε διεθνές επίπεδο όλο χρόνο να γνωρίσει ότι δεν ισχύει πια αυτό. Άρα δηλαδή πρέπει να έχουμε κατά νου τις επιπρόσθετες επιστημονικές γνώσεις που προκύπτουν ε, σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις της που δεν σταματούν σε εθνικά σύνορα ή σε συγκεκριμένους τομείς ε, της οικονομίας. Ε, κάθε άλλο από την κλιματική αλλαγή πλήττονται πάρα πολλοί τομείς της οικονομίας. Αυτή τη στιγμή συζητάει ένα ε, διεθνές συμβούλιο για την ε, κλιματική αλλαγή τα θέματα και θα αναφέρει τα πορίσματά του πριν από την συνάντηση στη Λίμα. Πάντως, ε, από ό,τι φαίνεται, αν θέλουμε μία σωστή καλή συμφωνία στο Παρίσι, δηλαδή με τη συμμετοχή των μεγάλων οικονομιών, τότε θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή κατά 3,5 μέχρι 4 βαθμούς ε, Κελσίου. Ε, θα προβλέπεται ότι θα υπάρξει αύξηση της θερμοκρασίας κατά 4 βαθμούς Κελσίου ε, έτσι λοιπόν σε σύντομο χρονικό διάστημα και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να, στα συμπεράσματα του να αναφέρει θέματα ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης, αλλά και αποτυπώματος άνθρακα. Θέλουμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού με όλες τις άλλες χώρες του κόσμου ε, θα κερδίσουν την, ε, τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστούμε πολύ για τις ε, παρατηρήσεις σας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσβλέπω σε καλή συνεργασία με τους και ηγητές για να καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο πραγματικά θα εκφράζει τις προτεραιότητες της ε, Επιτροπής μας. Και το κείμενο αυτό ε, πρέπει να σταλεί και στους ε, συναντέλφους της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Τώρα, προσωρινό χρονοδιάγραμμα. Διορία η Παρασκευή αυτής της εβδομάδας, 5 Σεπτεμβρίου, 12 η ώρα, για την κατάθεση τροπολογιών. Η ψηφοφορία θα γίνει στην Ήτρα ε, Δευτέρα 7 Οκτωβρίου. Στις 5 Νοεμβρίου θα γίνει η ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, μετά από ένα μήνα δηλαδή, και το όλο θέμα ε, θα πάει στο Στρασβούργο στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Πάρα πολύ ωραία, τελειώσαμε ακριβώς την ώρα μας, στις 6 ε, η ώρα. Αύριο όμως μην ξεχνάτε, στις 10 η ώρα έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εδώ το πρωί στις 9 θα συναντηθούμε για να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας και δεν θα έχουμε πάλι αναβολή για 10 ή 15 λεπτά. Θα ξεκινήσουμε ακριβώς 9. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.